Καλημέρα σας. Καταρχάς, ως συνήθως, να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τη συνεδρία των συντονιστών ε, που έγινε χθε. Και να σας τις ανακοινώσω, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνονται. Οι συγητές. Υπάρχει συμφωνία για την αναδιατύπωση του τίτλου για το ε, θέμα, το οποίο θα λέγεται «Έκθεση για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ε, έγινε μία συμφωνία καταρχάν και η έκθεση ε, θα γίνει με εισηγητές από το ECR και τους Πρασίνους. Ε, πρέπει να έχουμε την συνένεση της διάσκεψης των Προέδρων, αλλά έχουμε ονόματα εισηγητών. Παρακαλώ. Yes, I do have a point ναι, ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Αυτό γίνεται μόνο εάν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο του ομιλητή και μόνον. Ε, στο παρελθόν έχω διαμαρτυρηθεί για το τι γίνεται με το web streaming. Αν μιλάω όπως μιλάω τώρα και εσείς έχετε ανοιχτό το δικό σας το μικρόφωνο, αυτό που θα συμβεί είναι ότι η κάμερα δεν θα ξέρει τι να κάνει και ενώ μιλάω εγώ θα δείχνει εσάς. Επομένως τα λόγια μου θα βγαίνουν από το στόμα σας και μπορεί να μην σας αρέσει κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Βέβαια όλο αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Ε, για κάποιου που κάνουν προπαγάνδα που και θέλουν να του βλέπουν για πολλή ώρα, καλύτερα να μην του βλέπουν ποτέ. Ευχαριστούμε, θα το λάβουμε υπόψη. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ανακοίνωση. Βερολίνο. Έγκριση για την τροποποίηση των ημερομηνιών. Αρχικώς είχαμε προβλέψει τις 14 και 15 Φεβρουαρίου, αλλά επειδή δεν υπάρχουν συνεδριάσει κοινοβουλευτικέ στο Βερολίνο εκείνε τι ημέρε. Επομένω, ζητήσαμε να μεταφερθεί η συνεδρίαση για τι 19 και 20 Μαρτίου. Αυτό το νέο αίτημα θα πρέπει να το εξετάσουμε, να το εξετάσει και πάλι η διάσκεψη των Προέδρων δηλαδή, διότι είχε δοθεί έγκριση για την προηγούμενη ημερομηνία. Ε, δεν θεωρώ βέβαια ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει ο πρόεδρος και άλλα επτά μέλη, δύο από το ΕΛΚ, δύο από τους σοσιαλιστές και από εκεί και πέρα οι άλλες ομάδες ε, θα καθορίσουν τη συμμετοχή τους. Όσον αφορά τη γνωμοδότησή μου για τις δημογραφικές στατιστικές, επειδή μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλήξει σε μια συνένεση η οποία θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, Νομίζω ότι σήμερα δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε όπως προβλέπετε. Θα μπορούσαμε ίσως να ξανασυζητήσουμε τα προβλήματα. Ναι. Ε, θα δούμε βέβαια από εκεί και πέρα, αφού αποφασιστεί, θα υπάρξει μία αίτηση για έγκριση για μία ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για ένα νέο καθεστώς που προκύπτει από την ε, απόσχηση ε, ενός κράτους μέλους, εάν τέτοιο προκύψει. Ε, αυτά λοιπόν για τις ανακοινώσεις. Δεν βλέπω ενστάσεις και μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση για δύο κοινά ζητήματα, το καθεστώς και η χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Εδρυμάτων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου και την τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εις βάθος ε, αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, που μας είχε ήδη παρουσιάσει η κυρία Γεννάκου στις 26 Νοεμβρίου και τώρα πλέον είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες για τον ε, χρηματοοικονομικό κανονισμό. Η που της αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, αλλά εμείς ε, θα συντάξουμε τη γνωμοδότησή μας και θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς από την κυρία Γιαννάκου να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, επισημάνατε και ο ίδιος ότι είχαμε μια πρώτη συζήτηση ε, στην Επιτροπή μας πριν ακόμα μάλιστα να τεθεί η έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, εν τω μεταξύ υπήρξαν ορισμένες επαφές με τον Επίτροπο καθώς και την Προεδρία του Συμβουλίου και επίσης υπήρξε μία συνάντηση στην οποία ε, συζητήσαμε με την εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, και με την ε, παρουσία στελεχών από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ε, νομίζω αυτά μας έχουν δείξει έναν δρόμο για μια συνεννόηση που πρέπει να υπάρξει με όλες τις πλευρές. Και βέβαια αναμένεται να συζητήσουμε το ίδιο θέμα και με τη νέα Προεδρία, την Ιρλανδική Προεδρία. Είναι περιττό να επισημάνω ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι στοιχείο της δημοκρατικής ζωής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα αυτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχουν κάτω από ένα καθεστώς ε, το οποίο δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή ε, στην Ένωση, όταν μάλιστα τα ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον ένα βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καλωσορίζουμε νομίζω την πρόταση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Σεύκοβιτ που ήρθε σε συνέχεια της πρότασης που είχε γίνει με τη δική μου έκθεση και που αφορούσε στην αξιολόγηση της χρηματοδότησης των κομμάτων επί της εκθέσεως του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Θα σημειώσω ε, ότι με την παρούσα έκθεση που προτείνει και τον κανονισμό προτείνει η Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα λειτουργούν υπό την ομπρέλα του ευρωπαϊκού δικαίου, στα οποία αποδίδουμε πλέον νομικό στάτους. Οτιδήποτε δεν ορίζεται από τον κανονισμό, θα μπορεί να ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα πολιτικά κόμματα. Διότι θα μπορούν ελεύθερα να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η έκθεση δεν ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Δεν ζητούνται περισσότερα χρήματα. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό από όλες τις πλευρές ώστε να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και ιδιαίτερα με το χώρο των μίντια που παρακολουθεί τα έξοδα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τα κριτήρια αναγνώρισης ενός κόμματος γίνονται πιο σαφή. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρέπει να εκπροσωπείται στο 1 τέταρτο των κρατών μελών από ήδη υπάρχοντα κόμματα τα οποία έχουν εκλεγμένους βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια ή ευρωβουλευτές. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να είναι κόμματα σε εθνικό επίπεδο και ότι μπορεί να είναι επίσης ανεξάρτητοι βουλευτές που να είναι εκλεγμένοι. Έτσι διευρύνουμε τη βάση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος. Εγώ δεν έχω ε, αντίρρηση επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα δημοκρατικών διεργασιών και να διέπονται από τις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης. Τα κόμματα και τα πολιτικά τους ιδρύματα όπου ένα κόμμα μπορεί να έχει μόνο ένα πολιτικό ίδρυμα με τη θέση σε ισχύ του κανονισμού θα αποκτήσουν νομική οντότητα και θα αναγνωρίζονται υπό το δίκαιο της Ένωσης σε κάθε ένομη τάξη όλων των κρατών μελών. Για να λάβει χρηματοδότηση όμως ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν Ευρωβουλευτή. Άρα διαχωρίζεται η αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ως ευρωπαϊκών από την χρηματοδότηση η οποία απαιτεί την παρουσία ενός εκλεγμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην εσωτερική διαμόρφωση και στην κατάρτιση των εκλογικών ληστών πρέπει να λαμβάνετε φυσικά και να προωθείτε ισότητα των φύλων χωρίς αυτό να δημιουργεί δεσμευτική υποχρέωση ποσόστοσης, ωστόσο αποτελεί βασική αρχή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ετησίως θα διαπιστώνει ότι τα εγγεγραμμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά τους ιδρύματα πληρούν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο registry του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αμφισβητήσει την δημοκρατικότητα ενός κόμματος ή και να κάνει παράπονα απευθυνόμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια ομάδα σοφών, ε, την ονομάζουμε έτσι, τριών σοφών, που θα προέρχονται από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, που θα κρίνει το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ είχα κάνει μια ενδιάμεση πρόταση να είναι η Επιτροπή που ασχολείται με τα συνταγματικά θέματα, ε, η οποία θα μπορεί να δίνει μια γνώμη γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει μια τελικά πρόταση συνδυαστική δηλαδή να υπάρχει επιτροπή σοφών να έχει δικαίωμα όπως έχει η επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων να διοργανώσει ε, ακροάσεις και να δώσει τη γνώμη της και τελικώς υπάρχει και το ευρωπαϊκό δικαστήριο το οποίο θα μπορούσε να δώσει τελική και αδιαμφισβήτητη γνώμη. θα μπορούν τα κόμματα να μοιράζονται το 90% της χρηματοδότησης ανάλογα με το μέγεθος, τον αριθμό των ευρωβουλευτών που διαθέτουν. Ενώ το 10% θα είναι ίσο για όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Μέχρι τώρα αυτό είχε την ισορροπία 85% και 15%. Θα μπορούν να υποστηρίζουν εξατομικευμένες καμπάνιες μελών βουλευτών ή μελών εθνικών κομμάτων αλλά για θέματα που άπτονται των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μπορούν βέβαια τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα άμεσα συνδεδεμένα πολιτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν μέρος της χρηματοδότησής τους για δημοψηφίσματα, για καμπάνιες δημοψηφισμάτων όταν όμως αυτές άπτονται ευρωπαϊκών θεμάτων αντικειμένων για τα οποία έχουν τεθεί ερωτηματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, κύριε Πρόεδρε, το στάτους αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή, συμπληρωμένο και από τις δικές μας προτάσεις, ε, αλλά και από τις προτάσεις που ήρθαν από την Νομική Επιτροπή, οι οποίες δεν διαφέρουν καθόλου από τις δικές μας προτάσεις. Είδα δηλαδή με ιδιαίτερη χαρά ότι η έκθεση της Νομικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά η πρόταση δεν απέχει από τις δικές μας προτάσεις ε, μαζί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεννόηση με το Συμβούλιο το οποίο φαίνεται πως στην αρχή χωρίς να έχει τίποτα συγκεκριμένο που να το αμφισβητεί κατά κάποιο τρόπο από ό,τι πληροφορηθήκαμε έδειξε κάποια ανησυχία νομίζω όμως ότι με τη συζήτηση που γίνεται οι ανησυχίες αυτές έχουν διασκεδαστεί Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει και θα καταφέρουμε να έχουμε τελικά μία πρόταση ε, η οποία θα μπορεί να είναι και πρόταση όλων μας ε, για να δώσουμε υπόσταση στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η Ένωση πια έχει ιδία νομική προσωπικότητα και δεν δικαιολογείται τα ευρωπαϊκά κόμματα να παραμένουν υπό ένα ασαφές καθεστώς ε, διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης κλπ. Αυτό θα δώσει και ένα μήνυμα σοβαρότητας και κύριε Πρόεδρε θα δώσει και ένα μήνυμα στους εθνικούς χώρους ε, ότι όπως τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έτσι και τα εθνικά κόμματα θα πρέπει επίσης συνεχώς να εξυγχρονίζονται, να γίνονται όλο και πιο δημοκρατικά και να ανταποκρίνονται στις κοινέ μας επιδιώξεις και στο ευρωπαϊκό μας μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου. Νομίζω ότι πριν περάσουμε στη συζήτηση θα πρέπει να ακούσουμε και τον ε, άλλο συντάκτη τη γνωμοδότησης για τι χρηματοοικονομικές πτυχέ. Ο κύριος Γκερέρο έχει το λόγο. Συγγνώμη, διορθώνω. Η κυρία Γκουρμάη, ε, η οποία πρέπει να φύγει μετά, η αντιπρόεδρο, είχε ζητήσει αν μπορεί να παρέμβει αμέσω. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γκουρμάη και τη δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα το λόγο γιατί πιστεύω ότι ήμουν πολύ τυχερή που δούλεψα μαζί με τη Μαριέτα για το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά, ε, ήθελα απλώς να ευχαριστήσω και βεβαίως θα μιλήσει ο Γκερέρο μετά από μένα και θα ήθελα να πω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι πακέτο. Ε, να ευχαριστήσω λοιπόν τη Μαριέτα για την έκθεση αυτή πολύ κρίσιμη αποφασιστική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία γενικότερα χρειαζόμαστε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα τα οποία να είναι ικανά να ε, προωθήσουν το σεβασμό των βασικών θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών. δεν χρειάζεται νομίζω να θυμίσω ότι η Ευρώπη βιώνει μια κρίση. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες εν πλήρη διαφανία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κοινοί κανόνες για τη διαφάνεια και για το σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών. Όμως τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν δυναμικά και να αντιμετωπίζουν την πολιτική πραγματικότητα στο βαθμό λοιπόν που ε, κάποιες βασικές αρχές τηρούνται δεν θα πρέπει να υπερφορτώσουμε με κανόνες την όλη υπόθεση. Βεβαίως θέλουμε καθαρή χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ε, θέλουμε χρηματοδότηση η οποία ο, να ανταποκρίνεται ή να αντικατοπτρίζει αν θέλετε την υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών η να αντικατοπτριζει αν θελετε την υποστηριξη των ευρωπαιων πολιτων θα πρέπει να δίνονται κάποια χρήματα πριν από τις εκλογές στα κόμματα και θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος για τα κόμματα αυτά και τα ιδρύματα που θα καλούνται να ορίσουν το δικό τους καταστατικό, το δικό τους εσωτερικό κανονισμό κτλ. Άρα θα πρέπει να βοηθηθούν και σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, με αυτή την έννοια θα πρέπει γρήγορα να εγκριθεί ο κανονισμός ο οποίος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω για την ε, καταχώρηση, registration και για τις ποινές. Ε, μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να επεκφύγει των ευθυνών του ε, και θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, οργανώσουμε τα πράγματα έτσι ούτω ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παρακάμψης κάποιων βασικών αρχών. Τώρα για την αντικατάσταση των ο, σοφών από την ΑΦΚΟ ή δεν έχω μ, ε, τελική άποψη, αποκρισταλωμένη άποψη, αλλά ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια έξωθεν ανεξάρτητη αρχή, αν μπορώ να το πω έτσι. Τώρα για τη συμμετοχή στις εθνικές ε, καμπάνιες ε, δημοψηφισμάτων θέλουμε βεβαίως να συμμετέχουν όλες τις ευρωπαϊκές στις συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά πράγματα και η συγγήτρια ε, έχει την ε, ίδια άποψη ελπίζουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε μια καλή συζήτηση για τα θέματα αυτά και συγγνώμη που πήρα το λόγο από τον κύριο ε, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Γιαννάκου ευχαριστώ Ευχαριστώ κυρία Κουρμά για την παρέμβαση πάντοτε είσαστε ακριβείς και συγκεκριμένοι πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κεραίρο, βλέπω ότι υπάρχει θέμα διδικαστικό που θέτει ο συνάδελφος Σέφιν. Παρακαλώ. Ε, point of order. Επί της διαδικασίας, Πρόεδρε, και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπε πριν ο κύριος Άγνιο. Ε, φαίνεται ότι δεν μεταδιδόμεθα από το διαδίκτυο. Είναι κρίμα πρόεδρε αυτό. Ε, οπότε τουλάχιστον να στείλουμε μια τολή διαμαρτυρίας προς το Γενικό Διευθυντή διότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Βεβαίω, δίκαιο το έτοιμά σα και η διαμαρτυρία σα, να σπάζομαι, μου είπαν ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα λόγω έλλειψη αρκετών καναλιών διαθέσιμων. Αλλά βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση. Το ε, καταγράφουμε το αίτημά σα. Ο κύριο Κεράρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την τελευταία μας συνεδρίαση εδώ στην Επιτροπή ΑΦΚΟ συνέβησαν κάποια πράγματα που συνεπάγονται μία αλλαγή στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει δική μου γνωμοδότηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι βασικές αυτές αλλαγές έχουν ως εξή. Πρώτα απ' όλα αποφασίστηκε ότι ο εισηγητής για αυτή την ε, έκθεση, η αρμόδια επιτροπή αν θέλετε, είναι η Επιτροπή Προπολογισμού. Άρα η Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων καλείται να καταρτήσει γνωμοδότηση ώστε να έρθει να συμπληρώσει την έκθεση της Επιτροπής Προπολογισμών. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή Προπολογισμών σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε αποφάσισε να περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και η ε, έκθεση ακού πριν ξεκινήσει την εκπόνηση της έκθεσης για τον προσωπικό κανονισμό ε, η Επιτροπή Προπολογισμών. Άρα η έκθεση για το δημοσιογραφικό κανονισμό και η δική μου γνωμοδότηση, πάντοτε για τον προπολογισμό, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δικασία για την έκθεση Γιαννάκου για το γενικό καθεστώς, καταστατικό συγγνώμη, των ε, ε, πολιτικών κομμάτων. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβα, εκτός αν λανθάνω. Πιστεύω ότι είναι ορθά αυτά που λέω. Και η ίδια απόφαση ελήφθη ή λαμβάνεται και από το Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται ε, και να συζητά την έκθεση Γιαννάκου και το, στο αντίστοιχο τμήμα γενικές υποθέσεις, ενώ το θέμα του δημοσιονομικού ε, κανονισμού θα συζητηθεί αργότερα από την αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου και εφόσον εγκριθεί πρώτα η έκθεση Γιαννάκου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν έχει κανένα νόημα εγώ σήμερα να σας παρουσιάσω μια γνωμοδότηση με μια σειρά τροπολογιών. Όταν η έκθεση που θα συνοδεύσει πρέπει να περιμένει, δηλαδή πώς θα οριστούν στο καταστατικό τα δημοσιονομικά στοιχεία. Ξέρετε, αυτό οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ενό ε, Ισπανού φιλοσόφου, δεν όλοι οι Γερμανοί ε, οι φιλόσοφοι στον κόσμο, ο οποίο είπε ότι οι μάτες προσπάθειες οδηγούν στη μελαγχολία. Πράγματι δεν έχει νόημα να κάνουμε μάτες προσπάθειες όταν αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε πρώτα την έγκριση της έκθεσης ε, Γιαννάκου. Οπότε, λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα έγγραφο εργασία. Ε, ήδη μάλλον το είχα ε, παρουσιάσει την προηγούμενη συνεδρίαση και σήμερα έτοιμος να ζητήσουμε κάποιες τροπολογίες. Όμως θεωρώ ότι είναι μάταιη αυτή η προσπάθεια. Εν κατακλείδη. Ίσως να σας μπέρεψε λιγάκι, ίσως να μακρηγόρησα και να φλιάρισα λιγάκι. Πάντως, να τα ξαναπώ. Η αρμόδια επιτροπή για να εκπονήσει έκθεση για το δημοσιονομικό ε, ε, κανονισμό είναι η Επιτροπή Προπολογισμών. Αποφάσισε όμως αυτή η Επιτροπή να, να ολοκληρώσει πρώτα η Επιτροπή ΑΦΚΟ την έκθεση για να και μετά θα ξεκινήσει την εξέταση της έκθεσής της η Επιτροπή Προλογισμού. Άρα η δική μου γνωμοδότηση εξαρτάται από αυτή την έκθεση. Περιμένω λοιπόν και εγώ να υιοθετηθεί πρώτα απ' όλα η έκθεση για να... Λογικό δεν είναι. Ας περιμένουμε λοιπόν για να βάλουμε τα πράγματα μια σειρά. Άντρο από και πέρα οι συνάδελφοι θέλουν μια, κάποια πρώτη ιδέα των δικών μου απόψεων, θα μπορούσα να σας στείλω ηλεκτρονικά μέσω email τις τροπολογίες που έχω λάβει υπόψη, αν και θεωρώ ότι είναι μια μάταιη άσκηση, αφού πρώτα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης Γιαννάκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυρέρο. Πολύ λογικά αυτά που μας είπατε, λογική πρότασή σας. Ξέρετε και χθες υπήρξε συνάντηση ανάμεσα σε μένα και τον ε, πρέσβη, τον Ιρλανδό πρέσβη Μοντγκόμερη, που θα έχουμε την τιμή ε, να έχουμε επαφέ μαζί το επόμενο εξάμεινο και του έθεσα το θέμα του νομικού καθεστώτο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και του δημοσιονομικού κανονισμού. Και του ζήτησα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό και η Ιρλανδική Προεδρία σε αυτό το ζήτημα. Έτσι το λέω ε, ενημερωτικά. Ο κύριο Νταφ. Um, Πρόεδρε, συμφωνώ γενικά με το σύνολο την έκθεσης της Μαριέτας Γιαννάκου. Κάποια επιμέρους θέματα βέβαια χρήσουν περαιτέρω διευκρίνησης Παραδείγματο χάρη, ποιο είναι το νομικό καθεστώς αυτών των πολιτικών κομμάτων μετά την αναγνώρισή τους στον ευρωπαϊκό στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νόμου όπως είπε η συγγέτρια πρέπει αν κατάλαβα καλά να καταχωριστεί κάνει το κόμμα σε εθνικό σε κάποιο κράτος μέλος για λόγους φορολόγησης κτλ. Αλλά ποιο είναι ακριβώς το νομικό καθεστώς αυτών των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή θα ήθελα ας πούμε, να ξέρω το Βέλγιο ας πούμε τι θα κάνει τα περισσότερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα βρίσκονται στο Βέλγιο, θα αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του βελγικού νόμου. Τότε οι βελγικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αυτό πάντως. Και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του νομικού καθεστώτος των ευρωπαϊκών κομμάτων υπό ευρωπαϊκό δίκαιο και των άλλων πολιτικών κομμάτων υπό εθνικό δίκαιο για να μπορέσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε τις διαφορές πρέπει να είμαστε ακριβείς πρώτο αυτό δεύτερο δεν ενθουσιάζομαι με την ιδέα ότι τρία σοφά ανεξάρτητα και εξαιρετικά άτομα μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το νόμιμο ή το, το ορθό της λειτουργίας των πολιτικών αυτών κομμάτων. Ούτε πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι ο διαιτητής στη συγκεκριμένη περίπτωση. διότι έτσι ε, έτσι αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ελέγχονται θέλετε από την ίδια την πολιτική αρένα στην οποία ανήκουν εμείς εγώ θα προτιμούσα να έχουμε μια άλλη αρχή λίγο πιο μακριά από τα θεσμικά όργανα η οποία να ελέγχει τη λειτουργία αυτών των κομμάτων του, αυτού του, της νομοθετικής πράξης, του κανονισμού κτλ. Τρίτο, η, η ανάγκη είναι αλήθεια, ε, είναι είναι πραγματικά ανάγκη τα πολιτικά κόμματα, τα ευρωπαϊκά να έχουν έναν ευρωβουλευτή μέλος για να χρηματοδοτηθούν. είναι λίγο παράξενο η ύπαρξη ενό Ευρωβουλευτή να καθιστά ένα κόμμα χρηματοδοτήσιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι μπορούν να υπάρχουν και υπερεθνικά πολιτικά κόμματα που, των οποίων τα μέλη να ελέγχονται σε ε, επίπεδο περιφερειακό ας πούμε ε, και που ενδεχομένως να φιλοδοξούν να γίνουν ευρωβουλευτές αλλά δεν είναι ευρωβουλευτές λοιπόν πρέπει να είμαστε λιγάκι ρεαλιστές νομίζω στην προσέγγιση μας Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε την, να ενδυναμώσουμε αν θέλετε διάσταση των, την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών θέλουμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν οπότε αυτό με τον το, με, το κομμάτι με τον Ευρωβουλευτή είναι μάλλον αντιπαραγωγικό. Τέλος, για τα όρια στις δαπάνες. Το κείμενο το αφήνει αυτό στην εθνική ευχέρεια το να τεθούν όρια στις δαπάνες. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν χώρες που, όπου δεν υπάρχουν όρια στις δαπάνες για τις προεκλογικές εκστρατείες. Ε, υπάρχουν και άλλα που είναι πολύ αυστηρά. Για να είμαστε λοιπόν σωστοί θα πρέπει να βάλουμε οροφές και μέγιστα για τις ε, δαπάνες ε, για τις εκστρατείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω φιλανδικά σήμερα. Ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι μια σημαντική έκθεση. Έρχεται η κατάλληλη στιγμή. Έκανε πολύ καλή δουλειά η συγγήτρια και την ευχαριστούμε για αυτό. Θα ήθελα όμως να κάνω με τη σειρά μου κάποια σχόλια. Όπως είπε και ο κύριος Νταφ, σχετικά με την παρακολούθηση και ποιος θα κάνει αυτή την παρακολούθηση για το κατά πόσον ε, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα φέρνουν εις πέρας ε, τους στόχους τους και τις αρχές ε, που δηλώνουν τα διέπουν, συμφωνώ με τον Άντριο. Δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός φορέας, αυτός που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε καν η Επιτροπή μας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε απόλυτα ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι στην μια τέτοια αξιολόγηση ενός ε, φορέα που λειτουργεί, αν θέλετε, ανταγωνιστικά ε, σε σχέση με εμάς. Δεν είναι μια δραστηριότητα ε, που εμπίπτει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια καθαρά νομική δραστηριότητα, ένα δικαστήριο δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναλάβουν αυτό το ρόλο, όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γενικότερα, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά γενικότερα, κατά τις αλλαγές ε, των κανόνων του συγχρονισμού στο μέλλον, θα έλεγα ότι το εφαλτήριο πάνω της σκέψης μας πρέπει να είναι η νομοθετική εξουσία που έχει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι νομοθέτης. Δεν μπορούμε να ζητούμε το Κοινοβούλιο να φέρει πέρας εκτελεστικά καθήκοντα. νομικά καθήκοντα, αν θέλετε. Διαφωνώ με κάτι τέτοιο. Πάντως, σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας δίνει ενοριστικό κείμενο, ενοριστική λύση και Ούτε την τροπολογία μπορώ να την υπερψηφίσω. Τώρα κάποια άλλα σημεία που θα ήθελα να θίξω. Σχετικά με μια διάταξη για τη φορολόγηση. Δεν θέλω ότι δικαιολογείται μια τέτοια μνήμα. Καλό είναι να μείνει η φορολόγηση εκτός. Επίσης, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων. και κατάλληλη χρήση τους. Πρέπει να το δούμε πιστεύω πιο προσεκτικά αυτό. Κατά πόσο δηλαδή οι που προτείνονται είναι οι πλέον ορθοί ή πως είναι και πολύ υπεροριστικοί σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες και την παρακολούθηση και ελέγχο της χρήσης των κονδυλίων για τις εκστρατείες. Ποιος θα έχει διαφορετική φορή από χώρα σε χώρα. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί και να κριθεί σε εθνικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι οι πολιτικές της διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα υπάρχουν ε, σημαντικέ διαφορέ. Οπότε πιστεύω είναι κάτι που πρέπει να κρυθεί σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Γιατριμέχη. Καλό του συναδέλφου πάντω να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Σόλτ που πρέπει να μας εγκαταλείψει στις 10. Οπότε, να του δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που έδειξαν κατανόηση. Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε πανταχού παρόντες εδώ. Για τρία θέματα θα ήθελα να μιλήσω. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ακριβώς θίγει το ζήτημα πώς ε, θέλουμε να... Ε, πώς με βάση της ελευθερίας του συναθήριζεστε ε, που θέλουμε να γίνεται σεβαστή σε ολόκληρη την Ευρώπη πώς ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε σε τελευταία ανάλυση των πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όσο διαφανείς όσο πιο διαφανής γίνεται. Ε, όπως είπε και η κυρία Γκουρμάη, θα πρέπει το κείμενο να είναι ξεκάθαρο, σαφές, διαφανές, για να καταλαβαίνουν όλοι, όλοι οι πολίτες πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ε, και ε, πώς πρέπει να αντιδράσουν και εκείνοι. Και εδώ θα ήθελα δυστυχώς να πω και λυπάμαι πάρα πολύ που η κυρία Γιαννάκου δεν είχε το θάρρος να ε, πάει πιο πέρα. Βεβαίως τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι αυτόνομα, να έχουν ένα νομικό καθεστώς υπό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμως ξαφνικά υπάρχει η ανάγκη καταχώρησης σε ένα registry εθνικό βέλγικο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Αυτό είναι που δημιουργεί τη δυσκολία. Εμείς σαν κοινοβούλιο και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω και τη γνώμη της εισηγήτριας εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτόνομο νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ναι, και το, ε, ε, από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι αν, ποιος αναγνωρίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ωραία είναι όμως πολύ ασαφές το κείμενο η Ολομέλεια δηλαδή η Ολομέλεια θα ασχοληθεί με την αναγνώριση Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος ή η μια επιτροπή σοφών. Δεν είναι τόσο διαφανή τα πράγματα, δεν είναι τόσο κατανοητά για τον πολίτη. Και επειδή εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην δυσπιστεί προς εμάς ή προς τα πολιτικά κόμματα ο πολίτης, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Πρέπει να γίνει λίγο παραπάνω δουλειά όσον αφορά την ακρίβεια και τη διαφάνεια εδώ. Τώρα, Επόμενο θέμα για την ισοτιμία. Ισοτιμία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που μοιραία βρίσκονται σε κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Εγώ νομίζω ότι οι τροπολογίες 28 και 29 που αναφέρονται στην κατανομή των πόρων ε, δεν ε, ε, είναι ε, αν θέλετε όσον αφορά την ισοδυναμία, την ισοτιμία των ευρωπαϊκών κομμάτων έχουμε μεγάλα και μικρά κόμματα μέχρι τώρα ε, έχουμε μια κάποια αναλογία 85-15 ε, με αυτή την έννοια τα μεγαλύτερα κόμματα παίρνουν περισσότερη χρηματοδότηση ε, τουλάχιστον ας μείνουμε στο status quo ή ας ε, βρούμε ένα καινούριο τρόπο αλλά πρέπει να διατηρηθεί μια σωστή αναλογία Ευχαριστούμε κύριε Σόλτς ο κύριος Άγνη τώρα Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τα μέλη της Επιτροπής να κοιταχτούν στον καθρέφτη κατάματα και να σκεφτούν κατά πόσον έχουμε εντολή για να συζητούμε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θυμάμαι το 2009 να μας έλεγε ο κόσμος ότι ναι, ότι θα πρέπει να έχουμε αυτά τα πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, θα πρέπει να τα κάνουμε και εμείς ως ευρωβουλευτές θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη. Δεν θυμάμαι καθόλου κάτι τέτοιο έχουμε μια διαδικασία που πάει από πάνω προ τα κάτω. Οι Ευρωβουλευτέ έρχονται εδώ και λένε θα έχουμε πολιτικά κόμματα. Κανονικά θα έπρεπε να ισχύει το αντίστροφα. Ο κόσμο θα έπρεπε να συναντιέται στι παπ και στα εστιατόρια και να λέει δεν μα αρέσουν τα πράγματα όπω τα λέτε εσεί και θα δημιουργήσουμε μια ομάδα, ένα κόμμα για να αλλάξουμε τα πράγματα και θα είναι αυτοχρωματοδοτήματα. Εγώ ανήκω σε ένα τέτοιο κόμμα στο UKIP και δεν μα χρηματοδοτεί κανεί άλλο εκτό από εμά και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι πραγματικά μπαίνετε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και προσέξτε, λέμε ότι είναι άδικο να υπάρχουν τα κριτήρια του να είναι κάποιος μέλος ε, σε αυτό το ε, ε, πολιτικό κόμμα. Μάλλον για να υπάρχει πολιτικό κόμμα να υπάρχει ένας ευρωβουλευτής εδώ. Εάν λοιπόν μια πολιτική ομάδα δεν μπορεί να έχει αρκετή στήριξη για να έχει έναν ευρωβουλευτή, είναι σωστό να λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πληρωμένη εκπροσώπηση στην Ευρώπη. Με ανησυχεί λίγο αυτό το πράγμα. Στο το πάμε στην, στα άκρα, να δούμε ένα πολύ ακραίο παράδειγμα. Έστω ότι κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν το δημόσιο απαγχωνισμό. Δεν υπάρχει πολιτική στήριξη τη χώρα του, αλλά επειδή κάποιο άλλο στην Ευρώπη υπάρχει, ε, έχει, υπάρχει μια περιοχή που του στηρίζει περισσότερο, λέμε ότι υπάρχει δημοκρατική εντολή γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι ο Άντριου Νταφ ε, έχει κατά νου κάτι το οποίο καταλαβαίνω. Φοβάται ότι οι φιλελεύθεροι θα χάσουν τις ε, πολλές ψήφους στις επόμενες εκλογές και θέλουν να έχουν μια κάποια στήριξη. Δεν θα πρέπει όμως να προχωρούμε έτσι. Τώρα, ο προπολογισμό. Όλοι ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί διακαώ περισσότερο προπολογισμό και τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένοι να του τα δώσουν. Σα παρακαλώ λοιπόν, δεν είμαστε ο κατάλληλο χώρο να αποφασίσουμε τέτοια πράγματα. Ο κύριο Μπρόντ. Ναι. Τα πολιτικά κόμματα εκφύσεως είναι εθελοντικοί αυτόνομοι οργανισμοί που θεμελιώνονται από πρωτοβουλία των ιδρυτών τους και όχι από το κράτος. Ε, και μάλιστα το, κρέο, το κράτος να αναλάμβει αν η πρωτοβουλία είναι κάτι περαιτό. Το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει κάτι τέτοιο και παρευστρεί σε μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ομάδας πολιτών. Υπάρχουν λοιπόν δύο πιθανά προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να υπερκεράσουν τα πολιτικά κόμματα. Καταρχάς ε, τα κριτήρια σύστασής τους και επίσης τα κριτήρια για την ε, καταχώρησή τους. Εάν η διαδικασία καταχώρησης γίνεται απλώς και μόνον για να μην έχουμε κόμματα με το ίδιο όνομα, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η ικανότητα να καθυστερήσουμε την καταχώρηση ή την αναγνώριση ενός πολιτικού κόμματος για οποιοδήποτε άλλο λόγο ε, είναι κάτι ε, διαστραμμένο και έχει σχέση με την ε, Σοβιετική Επιτροπή Εκλογών. Αυτοί που ανήκουν σε ένα κόμμα έχουν κοινά συμφέροντα, κοινά ενδιαφέροντα αν ένα κράτος ή ένας υπερεθνικός οργανισμός λέει στα πολιτικά κόμματα τι αρχές θα πρέπει να προσυπογράφουν, είναι αυταρχικό. Και ακόμα και αν είναι καλή η πρόθεση και πάλι είμαστε απολυταρχικό καθεστώς σε αυτή την περίπτωση. Άκουσα τι είπαν ο κύριος Ντάφ και η κυρία Γιατενμάκη. Εκτιμώ τα όσα είπαν ότι αυτός ο οποίος λαμβάνει την απόφαση για την καταχώρηση και τη χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος φορέας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα κριτήρια θα έχουν ήδη καθοριστεί από πολιτικούς εδώ και στο Συμβούλιο που χώνουν τη μύτη τους παντού και νομίζω ότι υπάρχει μία παροχημένη έκφραση μεν, αλλά θα την ε, επαναλάβω ότι αυτός που πληρώνει αποφασίζει και τι μουσική θα παίξουμε. Λοιπόν, αυτό ε, ουσιαστικά διέπει τα πολιτικά κόμματα και ουσιαστικά έχουμε πολιτικά κόμματα στην υπηρεσία του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να προτείνω και εγώ κάτι που ήδη ελέγχθη να πω ότι τελικά το εκείνο που ε, μας ενδιαφέρει εδώ είναι το πώς γίνεται η χρηματοδότηση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι λίγο παράξενη και είναι λίγο ανισόρροπη με την έννοια ότι σε ορισμένα μέρη μπαίνει σε υπερβολικές λεπτομέρειες, σε ορισμένα άλλα είναι πολύ θολή. γιατί η δημοκρατία είναι αρκετά θολή αν θέλετε η έκθεση για Γι' αυτό εγώ έχω πρόβλημα. Από την άλλη μεριά βέβαια με για τη χρηματοδότηση μπαίνει σε αρκετές λεπτομέρειες ο κύριο Νταφ λέει δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες ε, είναι λοιπόν λίγο ανισομερή η έκθεση αυτή αυτό θα η πρόταση που έγινε από τη Κομισιόν ε, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία και γι' αυτό αποκτά πάρα πολύ μεγάλη σημασία η έκθεση της ε, συναδέλφου κυρία Γιαννάκου γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε να κάνουμε μια μελέτη για τα πολιτικά κόμματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια μελέτη η οποία να μπορεί να, την οποία να μπορεί να διαβάσει και ο πολίτης και να μπορούν λοιπόν να, ενημερώνουν, να ενημερωθούν όλοι για το τι προτιθέμεθα να κάνουμε στις Βρυξέλλες. Ε, άλλο θέμα τώρα. Ποιο είναι το νομικό στάτους των πολιτικών ε, κομμάτων. Πότε μια ομάδα γίνεται πολιτικό κόμμα και πότε χρηματοδοτείται. Κατά τη δικιά μου την άποψη δεν μπορεί να θεωρείται ε, πολιτικό κόμμα μια ομάδα μο, α, μόνο αν έχει μέλος έναν ευρωλευτή το θέμα είναι αν το, η συγκεκριμένη ομάδα θέλει να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία με ευρωπαϊκή και διαστάσεις και να λάβει μέρος αν θέλετε και στις ευρωπαϊκές εκλογές ε, δεν μπορεί να ορίζεται αυτό από το αν έχει μέλος ευρωβουλευτή ή όχι. Ε, μας ενδιαφέρει μια ομάδα πολιτική να έχει ε, ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα ευρωπαϊκά πράγματα και από εκεί και πέρα ποιος βεβαίως θα έχει κάνει τον έλεγχο για τα κόμματα κατά πόσον ισχύουν κάτι τέτοια πράγματα. Εμένα μου φαίνεται λιγάκι γελίο να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει για το κατά πόσον ένα κόμμα είναι κόμμα. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αυτά τα ε, ε, υπάρχουν άλλα κριτήρια δημοκρατική ε, δημοκρατικές δομές κίνηση από τη βάση προς τα, προς τα πάνω ε, τέτοιου είδους κριτήρια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το άλλο θέμα, όπως σας είπα, πέρα από το νομικό στάτους, είναι πώς χρηματοδοτούνται τα κόμματα. Εάν τα κόμματα είναι έτσι όπως φαντάζομαι εγώ, με δημοκρατικές δομές κλπ. κλπ άσχετα από το αν έχουν ή δεν έχουν ε, ευρωβουλευτές, ε, χρηματοδοτούνται ανάλογα από, με το μέγεθός τους που δεν είναι λόγο πρέπει να δεχθούμε δομές από εκ των άνω προς τα κάτω όχι από τη βάση προς τα πάνω τι να σας πω τώρα ποιος θα κάνει τον έλεγχο ο Όλαφ ή δεν ξέρω ποιος άλλος αυτές είναι διοικητικές βεβαίως λειτουργίες δεν με πειράζει, ας τις αναλάβει κάποιος φορέας ελέγχου, α, δεν ξέρω βέβαια αν ο, η Όλαφ είναι ο αρμόδιος φορέας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να μην γίνονται παρανομίες με την έννοια, μάλλον παρατυπίες θα έπρεπε να πω, να μην παρακάμπτονται κάποιες βασικές αρχές και αν έχουμε ορίσει το κόμμα με βασικά κριτήρια τις δημοκρατικές δομές ε, από τη βάση προς τα πάνω και τα λοιπά που είπα πριν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να ξαναελέγχονται από την ελεγκτική αρχή και αν δεν πληρούνται πλέον δεν χρηματοδοτείται το κόμμα αυτό τώρα και κάτι τι άλλο θα ήθελα να πω ο συνάδελφος Σούλτς είπε κάτι το οποίο δεν το θεωρώ σωστό. Τα κόμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται το εκείνο το οποίο σχετίζεται και η χρηματοδότηση πρέπει να σχετίζεται και με την στήριξη που έχουν σε κάποια χώρα ή κάπου στην Ευρώπη αν θέλετε τα κόμματα αυτά. Η στήριξη μετριάται όχι από, από δημοσκοπήσεις αλλά από ε, εκλογές από τις εκλογές άρα δεν πρέπει να βάζουμε οροφές αλλά θα πρέπει να βάζουμε κατόφλια το θέμα δεν είναι να πούμε 90-10 για να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο τους μεγάλους. Το θέμα είναι να πούμε 90-10 αλλά να έχουμε το κατόφλιο των 10 για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και τα μικρά κόμματα. Τώρα, έρχομαι σε λεπτομέρειες 18.3 λέει εκεί ότι δεν μπορούν τα α, πολιτικά κόμματα να λάβουν μέρος σε, σε δημοψηφίσματα για την Ευρώπη και τα λοιπά για το όνομα του Θεού τι είναι αυτή, ευνουχίζουμε τα κόμματα αυτά κατά το δοκούν θέλουμε τα κόμματα αυτά να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με την Ευρώπη. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για μια οδηγία η οποία ασχολείται με την α, ευεξία και την, ε, των ζώων. Μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουμε να τα βοηθήσουμε και αν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να βοηθήσουν στις τοπικές εκλογές να βοηθήσουν στις τοπικές εκλογές στη δική μου, στο δικό μου το Δήμο θα ήθελα πράγματι να έρθουν να βοηθήσουν κάποια ευρωπαϊκά κόμματα Είμαστε ένα πολιτικό σώμα γενικώ. Δεν μπορούμε ορισμένα κόμματα να, επιτρέ... να μην τους απαγορεύουμε να κάνουν ορισμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτικό όργανο αλλά ε, είναι νομοθετικό όργανο. Εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα. Δεν θα έπρεπε να ζητούμε νέους φορείς ή ακόμη και το ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ελέγχει ορισμένα πράγματα. Είναι νομοθέτης που φτιάχνει το πλαίσιο. Άλλοι είναι οι φορείς που θα ελέγξουν. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Έφνερ θα πάρει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά συζητούμε Εκτεν... Δεν, είναι... δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή. Γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που το ανέφερε και ο συνάδελφος Βίλαντ. Και το οποίο είναι σημαντικό. Πριν από 1,5 χρόνο ε, κάναμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό. Το συζητούμε το ε, θέμα αυτό και ο Βίλαν και ο Νταφ μίλησε ε, για το θέμα αυτό ή πιο ότι είναι νομικά απαραίτητο η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων να μην εξισούται ή με την αναγνώριση, καταχώρηση, registration των πολιτικών κομμάτων. Η χρηματοδότηση μπορεί να σχετίζεται με την επιτυχία και τη στήριξη ενός πολιτικού κόμματος, αλλά η καταχώρηση ε, ενός πολιτικού κόμματος δεν μπορεί να συνδέεται με την επιτυχία του και με τη στήριξή του το, θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να είναι ελεύθερα να εκφράσουν οποιαδήποτε άποψη είτε είναι δημοφιλής είτε όχι είναι τελείως άλλο πράγμα λοιπόν registration από την χρηματοδότηση και εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι κατά πόσον οι πολίτες, τα πολιτικά κόμματα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί την Ευρώπη συνειδητοποιήσουν ότι θέλουμε να είμαστε δίκαιοι να δημιουργήσουμε μία αρένα ε, αγώνα μεταξύ πολιτικών κομμάτων που μπορεί να είναι οτιδήποτε ε, να εκφράζουν οποιαδήποτε άποψη η πρόσβαση στην αρένα αυτή δεν μπορεί να περιορίζεται αλλά η χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να εξαρτάται από την επιτυχία. Η registration όμως δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Αν δηλαδή ο πολίτης σκεφτεί με αυτά που λέμε ότι με βάση αυτά που λέμε ότι δεν θέλουμε κάποια πολιτικά κόμματα, δεν θέλουμε κάποιες απόψεις να εκπροσωπούνται από πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη ο Θεός να μας βοηθήσει. Είναι κάτι που επουδενή λόγο θέλουμε να κάνουμε. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ επικίνδυνο να, μπορέ, να, να μπερδέψουμε εδώ τη registration με τη χρηματοδότηση. Για τη registration υπάρχουν τυπικά επίσημα κριτήρια, δεν ξέρω, ο αριθμός των ενώσεων, ο αριθμός των χωρών, ο, δημοκρατικές δομές ε, και τα λοιπά. Ε, αν υπάρχει βούληση να συμμετάξει ε, το κόμμα αυτό αυτό που θέλει να ε, γίνει κόμμα στις ευρωπαϊκές εκλογές ε, όπως είπε και ο Βίλαντ εδώ δεν είναι η registration δεν είναι πολιτική απόφαση είναι διοικητική απόφαση Μέχρι εδώ καλά, συμφωνώ με τον Βίλαντ. Από εκεί και πέρα όμως παίρνουν την εξουσία οι πολίτες και η χρηματοδότηση ανάλογα με την επιτυχία που έχει το κόμμα, ανάλογα με τη στήριξη που έχει από τους πολίτες δίνεται μετά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προ, προσέξτε το πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ ήδη έχουμε ετοιμάσει τις τροπολογίες αλλά ελπίζω να μην έχουμε διαφορετικές απόψεις και να μην τσακωθούμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή διότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να είναι ομόφωνη όσον αφορά το τι εστί Ευρωπαϊκή Δημοκρατία εδώ μιλάμε για πράγματα για τα οποία δεν έχουμε άμεσο συμφέρον εμείς. Δεν προσπαθούμε να περάσουμε τις δικές μας ιδέες. Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί για να μπορούν να εκφραστούν οι πολίτες. Τώρα, να η, συμμετοχή στα δημοψηφίσματα. Συγγνώμη, εδώ πού πρέπει να βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή, την κόκκινη γραμμή. Αν να υπάρχει κάποιο δημοψήφισμα με με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον τι γίνεται, απαγορεύεται τα κόμματα αυτά να κολλήσουν αφήσει ή να κάνουν κάτι. Συγγνώμη, δεν θέλουμε να συμμετάσχουν στην στη μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το ναι όχι ε, στην Ευρώπη για το ναι ή όχι ε, των δημοψηφισμάτων έχω αμφιβολίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην κόκκινη γραμμή να μην θα βάλουμε εδώ για να μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένα πράγματα σωστά στην πράξη. Τώρα για την κατανομή ε, κατόφλια, οροφές κτλ. Εδώ έχω διαφορετική άποψη από τους προλαλήσαντες. Καταλαβαίνω βέβαια τι είπαν. Ε, πιστεύω όμως ότι είναι απαραίτητο και σωστό ένα μέρος του πώς το ένα μέρος της χρηματοδότησης να πάει για τα λειτουργικά έξοδα αν θέλετε των κομμάτων και ουσιαστικά ε, τα λειτουργικά έξοδα είναι περίπου τα ίδια ε, για όλα τα κόμματα και μετά μπαίνει ο παράγοντας της επιτυχίας. Το 85-15 εγώ πιστεύω ότι είναι καλό ποσοστό, καλή αναλογία. Το 90-10 πάει λίγο πιο μακριά, αλλά τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν και επιφυλασσόμεθα να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Ε, ε, Καλώς. Ε, Απαντήστε στην κυρία Κουρμάη, παρακαλώ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Χίλια συγγνώμη. Δικό μου το σφάλμα. Δεν πρόσεχα λιγάκι και να, τι συμβαίνει. Και τώρα θα σας προσέχω απόλυτα, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι. Φυσικά την απάντηση θα δώσει η κυρία Γιαννάκου. Και αν από εκεί και πέρα ο κύριος Γκερέρο θέλει να τοποθετηθεί εκ νέου, με χαρά. Ίσως να δώσουμε πρώτο το λόγο ε, στον κύριο Γκερέρο για να κλείσει τη συζήτηση η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω σε σχέση με όσα είπα πριν πριν είπα ότι πρέπει να περιμένω πρώτα να εγκριθεί η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου για να δω τι συνέπειες θα έχει στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτή τη στιγμή και η Επιτροπή Προπολογισμών και η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να δούμε πώς η μεταρρύθμιση του ιστορικού κανονισμού θα επηρεάσει τα πράγματα και βεβαίως πρέπει να δω την έκθεση Γιαννάκου πρώτα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου, θέλω να καταγράψω το εξή. Πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι μείζονο σημασία. Δεύτερον, πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα πριν ληφθούν οι αποφάσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά να προσθέσω κάτι ακόμη. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκά και όχι απλά να είναι το άθροισμα εθνικών πολιτικών κομμάτων που εκφύσεως βλέπουν την Ευρώπη ως τον τόπο όπου μπορούν να περασπιστούν τα εθνικά του συμφέροντα. Όχι, το αντίθετο θέλουμε κόμματα που πραγματικά να έχουν την πρόθεση να εργαστούν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ε, υλοποίηση του μεγάλου ευρωπαϊκού οράματος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα απλό αριθμητικό άθροισμα των κομμάτων, αλλά για μια σύνθεση απόψε. Με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε τα πράγματα. Και ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στον εκλογικό, α, τις εκλογές, αν θέλετε, με όλες τις άλλες λειτουργίες. Γιατί τα κόμματα δεν έχουν μόνο το ρόλο να στηρίξουν τους υποψήφιους εκλογές και να εκδίσουν εκλογές, αλλά έχουν άλλο καθήκον να στηρίξουν ε, μια δημοκρατία, να παρουσιάσουν προγράμματα και να προσπαθήσουν να πείσουν την κοινή γνώμη για τις θέσεις τους. Αυτό είναι ε, βασικό καθήκον των κομμάτων που διαφέρει βεβαίως αν και άλλο σημαντικό καθήκον είναι η στάση τους στι εκλογές και η εκλογική διαδικασία εν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεται πολύ ελευθερία στην ε, διαμόρφωση ε, ενό κόμματο και άλλο πράγμα ο δημοκρατικός μεν, αλλά έλεγχος κατά την εκλογική διαδικασία. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση συμβολιστή και θα σα υπενθυμίσω και ένα σεμινάριο που κάναμε για τα πολιτικά κόμματα. Και υπάρχουν τα πρακτικά. Δεν ξέρω, όπω είπε ο κύριο Βίλαντ, αν μπορώ να ζητήσω τη μετάφραση των πρακτικών αυτών σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω αν προβλέπετε από τους κανόνες. Θα ζητήσω πάντως να μεταφραστούν αυτά τα πρακτικά. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. Πάλι λάθος το όνομά σα. Ελπίζω να μην αρχίζουν να, να με βλέπουν με υποψία οι συνάδελφοι. κυρία Γιαννάκο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερο την κυρία Γκουρμάη για τις πολύ α, α, επικοδομητικές και κολακευτικές θα έλεγα, <clears throat> τα κολακευτικά σχόλιά της Εξ όσων αντελήφθη τους συναδέλφους απασχολεί η υπόθεση του πώς θα αναφέρεται και θα θεωρείται ένα κόμμα ότι είναι ευρωπαϊκό, δηλαδή αυτό το registration και πώς θα γίνεται και τους απασχολεί το τμήμα εκείνο των παραπώνων που μπορεί να κάνει ένας πολίτης ή μια οργάνωση και ποιος θα κρίνει αν τα κόμματα αυτά είναι ε, δημοκρατικά ή όχι και γι' αυτό είπα ότι ίσως ένας συνδυασμός ε, μιας γνώμης της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων με την Επιτροπή αυτή των Σοφών ε, που θέλει η Κομισιόν και ίσως τελικά μια απεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το Κοινοβούλιο γιατί δεν είναι εύκολο και σε πολιτικό επίπεδο να κρίνουν πολιτική κόμμα που είναι σε ένα κόμμα ένα άλλο κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται θέμα αξιοπιστίας. Ε, θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα αυτό. Δηλαδή εν τέλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να λύσει τις αμφισβητήσεις για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα στους συναδέλφους που ανέφεραν ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα ε, θα πω ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία είναι στο Βέλγιο, είναι στις Βρυξέλλες και λειτουργούν ως διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, πληρώνουν τεράστιους φόρους κτλ. Δηλαδή δεν ερχόμαστε για πρώτη φορά να θεσμοθετήσουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν και χρηματοδοτούνται. Και επομένως πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες. Τώρα το θέμα της νομικής προσωπικότητας είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που ανέφερε ο Άντριου. Ε, ό,τι δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό ο κανονισμός είναι υποχρεωτικός για τα κράτη-μέλη. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό θα ρυθμίζεται από το κράτος μέλος αν το κόμμα εγκατασταθεί στη χώρα αυτή. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία εγκατάσταση. Μπορεί ένα κόμμα αν θέλει να εγκατασταθεί στη Μαδρίτη ή στο Βερολίνο. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό θα το ρυθμίζει ο νόμος της Γερμανίας ή της Ισπανίας και νομίζω αυτό είναι δίκαιο και σωστό. Το ίδιο ισχύει και για ένα πλήθος ε, οδηγιών και κανονισμών που υπάρχουν και που συνομοθετεί το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι τίποτα περίεργο. Είναι η συνήθις νομοθετική πρακτική η οποία υπάρχει. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας ε, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν νομοθεσίες για τα εθνικά κόμματα αλλά αυτό είναι μια τελείως άλλη υπόθεση. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα οφείλουν να έχουν συγκεκριμένο καθεστώς, το έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο επανειλημμένα και βέβαια οφείλουν κυρίως να προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τώρα, εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν την προώθηση και την εξέλιξη της Ευρώπης ε, και αυτές έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν μέσω κομμάτων και να λένε αυτά που θέλουν να λένε. Δεν εμποδίζει κανείς κανέναν ως προς το περιεχόμενο των ιδεών Εάν βέβαια υπάρξουν κόμματα τα οποία θα μεταχειρίζονται αντιδημοκρατικές πρακτικές τότε βεβαίως υπάρχει αντικείμενο το οποίο μπορεί να κριθεί ε, και νομίζω ότι έχουμε όλα τα μέσα και ως κοινοβούλιο και ως θεσμικά όργανα ε, έχουμε όλα τα μέσα στα χέρια μας για να μπορούμε να κρίνουμε ε, παρόμοιες καταστάσεις. Τώρα το θέμα που εθίγει ως προς το φορολογικό αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ό,τι δεν προβλεφθεί από τον κανονισμό μπορεί να το ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητα σε όλα τα ζητήματα. Επομένως δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Μας ενδιαφέρει όμως τα κόμματα αυτά να υπηρετούν όσο το δυνατόν α, τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και ταυτόχρονα να διέπονται από διαφάνεια. Και εφόσον διαθέτουμε τα μέσα για να ελέγξουμε τη διαφάνεια των διαφόρων πράξεων νομίζω ότι αυτό είναι πολύ απλό. Κατά τα άλλα όπως σας είπα θέμα αύξησης της χρηματοδότησης δεν τίθεται. Αν θέλετε τίθεται θέμα νομιμοποίησης σωστού ευρωπαϊκού στάτους και νομικής προσωπικότητας των κομμάτων πράγμα που θα τους προσδώσει κύρος και ιδιαίτερη αξία και σεβασμό στα κράτη-μέλη διότι τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα αλλά δεν έχουν νομική ουσιαστική προσωπικότητα. Μία νομική προσωπικότητα θα τους προσδώσει μια ιδιαίτερη αξία ε, μέσα στο χώρο των κρατών μελών και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και η δυνατότητά τους να γίνονται μέλη αυτών των κομμάτων ε, και να λαμβάνουν γνώση από τα κόμματα αυτά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδέα οι ευρωπαίοι πολίτες ποιος αποφασίζει τι και για ποιο λόγο. Σε καμία από τις χώρες μας. Αν θέλετε στη δική μου χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος έμαθε πάρα πολλά πράγματα για την Ευρώπη στα τελευταία τρία χρόνια. Αλλά οι περισσότεροι πολίτες στην Ευρώπη τι ξέρουν για το ποιος παίρνει τις αποφάσεις, πώς παίρνει τις αποφάσεις, τι γίνεται. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν και αυτά ένα ρόλο στο να επικοινωνήσουν με τους πολίτες και να δείξουν στους πολίτες ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Συνήθως οι κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι ό,τι έρχεται από τις Βρυξέλλες είναι κακό και ό,τι έρχεται από την πρωτεύουσα και από τις κυβερνήσεις είναι καλό. Αυτό μπορούν να το εξισορροπήσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Και νομίζω πως την αξία των κομμάτων με ένα σαφές νομικό καθεστώς θα τη βλέπουμε στο βάθος του χρόνου να είναι όλο και ισχυρότερη κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις όλων των μελών σε τροπολογίες που θα κάνω η ίδια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν μια κοινή άποψη πρώτον εμείς μέσα στην Επιτροπή τη δική μας και δεύτερον να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ ειλικρινά κυρία Γιαννάκου για τα όσα κάνατε πολύ σημαντική δουλειά σας, όπως είναι και πολύ σημαντική συζήτηση που έγινε και που θα ξαναγίνει να δούμε πότε. Προθεσμία για την κατάθεση προ... τροπολογιών για τις 17 Ιανουαρίου, ενώ ψηφοφορίες που θα μπορούσε να γίνει στις 19 Φεβρουαρίου. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά, είναι η αλήθεια για το θέμα αυτό, αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις... σε αυτή τη θητεία τουλάχιστον, πρέπει ε, να ακολουθήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 11 για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Αποφασίσαμε ήδη να μην ψηφίσουμε το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να κάνουμε μια νέα ανταλλαγή απόψεων ε, για το θέμα αυτό, όπου δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, υπάρχουν αμφισβητούμενα σημεία, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, ε, κατά την άποψή μου είναι δύο. Το πρώτο και πιο σημαντικό από όλα αφορά τις επιπτώσεις των δημογραφικών στατιστικών οι επιπτώσεις των δημογραφικών στατιστικών στα θεσμικά όργανα. Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο, η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν τα στατιστικά στοιχεία έχουν απλώς ε, επιπτώσεις ε, για λόγους γνώσης που μπορεί να έχουν και κάποια επιρροή σε κάποιους τομείς όταν επιχειρηματολογούμε και σκεφτόμαστε και πολιτικά ζητήματα ή αν μπορούν να έχουν και ε, επιρροή στα θεσμικά όργανα και ποια επιρροή σε αυτή την περίπτωση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Αν βασιζόμαστε απλώς και μόνο στα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, στη Eurostat, ή αν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία. Αν λαμβάνεται υπόψη η υπηκότητα, ε, η διαμονή, ε, το θέμα της παραμονής. Ε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίε κατά την άποψή μου, γιατί στα διάφορα κράτη-μέλη η έννοια της δια, παραμονής, της διαμονής δεν είναι ίδια. Ε, στην Ιταλία, για παράδειγμα, είναι η συνήθις κατοικία. Όποιο λοιπόν διαμένει κάπου έχει το κέντρο των συμφερόντων του και των επιχειρήσεών του εκεί. Υπάρχουν όμως κάποιες τροπολογίε που προσπαθούν να ορίσουν τη διαμονή με κάπω διαφορετικό τρόπο, πιο περίπλοκο, ε, πιο ιστορικό σε κάποιε περιπτώσει και γίνεται και μια σύγχυση ε, του όρου τη διαμονή. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο περισσότερο τα θέματα αυτά, αν θέλουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενό μας και σίγουρα θα πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Να υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία που να καλύπτει όλες σας τις ανησυχίες. Αυτή τη, ε, τη φορά πραγματικά δεν θα πω κυρία Γιαννάκου, έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως επειδή είμαι πολύ κοντά σας, ε, γι' αυτό κάνετε συνέχεια λάθος. Δεν θέλω να πω ότι είμαι νεότερη, δεν ξέρετε κανείς ποτέ βέβαια. Λοιπόν, για τα ευρωπαϊκά δημογραφικά στατιστικά. Καταρχάς, να συνεχίσω από το σχόλιο του Προέδρου. Νομίζω ότι καλή ήταν η απόφαση να αναβάλουμε την ψηφοφορία για να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε και να σκεφτούμε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση η συλλογή ακριβών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για τα δημογραφικά στοιχεία στην ε, Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά για το η χάραξη πολιτικής και την ε, ε, αξιολόγηση της συνεργής είναι ζωτική σημασίας και επίσης άπτεται ευαίσθητων θεμάτων, ιδίως σε χώρες και περιφέρειες με υψηλό ποσοστό οικονομικής μετανάστευσης και μετακίνησης. Αυτή η αύξηση λοιπόν στη μετακίνηση των πολιτών ε, διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης ε, που έχουμε συζητήσει επανελειμμένως και πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάποιων χωρών μελών. Από ό,τι βλέπουμε, τα στοιχεία αυτά θα έχουν και επιπτώσεις στην εκπροσώπηση των κρατών μελών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως στο Συμβούλιο. Εάν λοιπόν πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος η συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη μέθοδο συλλογής και να λάβουμε υπόψη και τι πολιτικές επιπτώσεις υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταρκόφσκι. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα, γιατί έχουμε συζητήσει όλες τις πτυχές του ζητήματος την προηγούμενη φορά. Να σας πω ότι είχαμε όμως δύο συμβιβαστικές προτάσεις επιτόπιτες και νομίζω ότι η ε, πρόταση του κυρίου Καζίνη ήταν σαφέστερη. Ξέρω ότι οι φιλελεύθεροι φίλοι μου θέλουν να καταλήξουν σε ένα καλό συμβιβασμό και οδεύουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε μεν με το πνεύμα, αλλά κατά την άποψή μου δημιουργείται μια κάποια σύγχυση με την ε, συμβαστική τροπολογία αυτή. Γνωρίζουμε όλα τα επιχειρήματα και το πιο σημαντικό είναι ότι λέμε ότι τα δικαιώματα της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων ε, είναι συγκεκριμένα, ιδίως όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Δεν έχουμε αποκλίνουσες απόψει. Απλώς νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι να ε, καθίσουμε κάτω όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις δύο συμβιβαστικές τροπολογίες, ίσως με κάτι εγκύτερο στην ε, τροπολογία του Προέδρου του κ. Καζίνη. Ε, γνωρίζουμε όλα τα επιχειρήματα και θα μπορέσουμε ίσως να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Σάκνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να, άλλη μια ευκαιρία να κερδίσουμε χρήματα. Αυτές οι στατιστικές θα κοστίσουν πολλά χρήματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε, να κάνουμε τη συλλογή αυτή των στατιστικών. Στη χώρα μου, ε, λόγω της μεγάλης εισόδου μεταναστών, ε, τα στατιστικά στοιχεία έχουν μπερδευτεί Κανείς όμως δεν έχει σωστά στοιχεία και δεν έχει σωστά στοιχεία στη χώρα μας λοιπόν επειδή μπερδεύονται τα πράγματα λόγω των μεταναστών που κάθε ώρα και στιγμή έρχονται στα σύνορά μας. Έχουμε χάσει τον έλεγχο. Ερώτηση λοιπόν πόσο αξιόπιστα είναι τα στοιχεία αυτά ε, και πόσο... Ε, και υπάρχει και το ενδεχόμενο ε, πραγματική σύγχυση. Βέβαια ο Ούγγρος συνάδελφος δεν βρίσκεται εδώ. Δεν ξέρω, θα ήθελα να τον ρωτήσω αν ήταν εδώ. Αυτοί που ζουν στην Τρανσιλβανία ε, είναι στην Ουγγαρία ή στη Ρουμανία πού βρίσκονται, πώς υπολογίζονται και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία. Παράδειγμα, η Ελλάδα ήθελε να μπει στην Ευρωζώνη. Χρησιμοποίησε για, με ένα αλφα τρόπο τα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν ε, παραπλάνησης μέσω αυτών των στοιχείων. Ε, λοιπόν, λάβετε υπόψη σε αυτό που είπα και ας γλιτώσουμε τα χρήματα που θα κοστίσει η συλλογή τους. Καταγράφουμε αυτές τις σκέψεις και θα προσπαθήσω και εγώ να βρω μία συμβαστική λύση με τις επαφές που θα έχω με όλους σας έως την επόμενη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου. Οπότε και θα σας πω πώς ε, θα προχωρήσουμε. Ελπίζω να πάμε και στην ψηφοφορία για να καταλήξουμε και σε κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. περάσουμε στο επόμενο σημείο. Και αυτό πολύ σημαντικό. στο επόμενο ε, σημείο έχουμε δύο συγκεκριτές ε, θεσμικά προβλήματα για μία ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο συγκριτέ, όπω είπα, Τρασκόφσκι και Γκουαλτιέρη. Σήμερα το κείμενο ε, είναι ένα έγγραφο εργασία στα αγγλικά και καλό του δύο συγκριτέ να μα το παρουσιάσουν. Κύριε Τρασκόφσκι, έχετε το λόγο. Ναι, αυτό το θέμα το έχουμε ξαναζητήσει δύο ή τρεις φορές ήδη και έχουμε καταστήσει σαφείς τις προθέσεις μας. Δεν θα ήθελα λοιπόν να αναμακρηγορήσω στην παρουσίασή μου, ιδίω εφόσον υπάρχει ένα έγγραφο ενώπιόν σας και ο στόχος μας ήταν να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο εργασίας για να μπορούμε να προετοιμαστούμε και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Προτιμήσαμε λοιπόν να μην υποβάλουμε ένα σχέδιο γνωμοδότηση, αλλά ένα έγγραφο εργασία. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο, για να διευκρινίσουμε τι έννοιε, όπω σα είπα και σε προηγούμενε περιπτώσει, ο να σαφέ δεν μιλάμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση και τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα. Θέλουμε να κινηθούμε ταυτοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνουν οι συνθήκες, να δούμε λοιπόν καλά τις συνθήκες και να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αφεληθούμε από αυτές για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το διάφορα γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι η ολοκλήρωση στα κράτη-μέλη γίνεται με διαφορετικό ρυθμό. Και πώς μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, με τη χρήση των συνθήκων, να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, αναρωτηθήκαμε ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση για να εμβαθύνουμε ε, σε αυτά τα ζητήματα με βάση την κείμενη συνθήκη. Βέβαια, ε, αυτό είναι σαν ένα κινούμενο στόχο. Γιατί κάποιε αποφάσει λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά συμβούλια και εκεί εμεί δεν έχουμε ουσιαστική συμμετοχή, ούτε έχουμε λόγο εκεί. Και επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων και μέχρι πού μπορούμε να πάμε χωρίς αλλαγή των συνδικών, γιατί καθώ κάποιε αποφάσει λαμβάνονται και είναι πολύ επίμαχε. Έπειτα, οι τρόποι με, τον οποίο, με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέγιστα το δυναμικό των συνδικών χωρίς αλλαγή τους. Σε πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταγράψαμε το γεγονός ότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, κάτι που δεν προσδοκούσε σε αυτό το βαθμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έπειτα και λίγα λόγια για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ώστε να εκπληρώσουμε και τους δικούς μας στόχους προτεραιότητες. Αν το δημοσιονομικό αυτό σύμφωνο γινόταν πραγματικότητα, κάτι που έγινε, να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να μην δημιουργήσει και να κατακαιρματισμό και νέους θεσμούς. Επειδή υπάρχει το ζήτημα της έκθεσης Tyson και πώς μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή. Ο Ρομπέρτο έκανε μια εξαιρετική γνωμοδότηση, χωρίς βεβαίως να έχουν ληφθεί υπόψη από την ΕΚΟΝ, αλλά πάνω σε αυτή την αγνώση μπορούμε να βασιστούμε και να ενισχύσουμε περισσότερο τη θέση μας. Τώρα για το μέλλον. Πρέπει να το σκεφτούμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Και φυσικά θέλουμε και τα σχόλιά σας και για όσα ανέφερα πριν. Και θα είναι πολλά τα σχόλια σας, αλλά πλέον, τα πλέον επίμαχα σημεία όπου πραγματικά είναι καλό να ενώσουμε τις προσπάθειές μας είναι το σημείο 5 ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε για το μέλλον, τι θέλουμε να κάνει η Ένωση λοιπόν στο ποτρό μέλλον. Και αυτό συνδέεται με το τελικό ερώτημα. Θέλουμε αλλαγή των συνθήκων και με ποιο τρόπο και τι θα θέλαμε να περιλαμβάνει νέα συνθήκη. Και το βασικό θέμα, το οδηγούν αν θέλετε σε αυτό το έγγραφο εργασία είναι ότι δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε την παγίδα που κάνουν πρόσφατα τα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουμε τέτοιες κατηγορίες. Θέλουμε και να δούμε αυτό το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα κοιτώντας προς το μέλλον. Η υπόθεση εργασίας ποια είναι όλα τα κράτη-μέλη είναι υπόκειτο στου κοινοτικού κανόνε, οι οποίοι διαφοροποιούνται σε θέματα οικονομική και νομισματική πολιτική και κατά πόσο οι πόροι που είναι διαθέσιμοι διαφοροποιούνται εξίσου. Θα πρέπει λοιπόν, κοιτώντα το μέλλον, να αναρωτηθούμε πώς θα γίνει αυτό πράξη. Και πάλι, αν δούμε το blueprint της Κομισιόν και τα επόμενα βήματα, με το paper του Βαν και όσα λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο, κατανοείται ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Βεβαίως, μας απασχολεί η μορφή της μελλοντική συνθήκης γιατί στο τέλος μιλούμε, στο έγγραφό μας μιλούμε για το ότι είμαστε πρώτον πυλών για την αλληλεγγύη της συνθήκης και εκεί υπάρχει ένα δίλημα. Από τη μία, θα πρέπει να δούμε συνταγματικά και θεσμικά ζητήματα, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, χωρίς να μπαίνουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Γιατί τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Εμείς και η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, δεν θέλουμε να μπαίνει μια επιτροπή στα χωράφια τη άλλη, ούτε επιστρέφουμε πολύ στα οικονομικά, αλλά ούτε εκείνοι να μπαίνουν στα θεσμικά ζητήματα. Άρα το ζήτημα είναι σε πόσο βάθο πρέπει να πούμε σε αυτά τα ζητήματα. Και ένα άλλο ερώτημα που τίθεται και συνδέεται με το πρώτο, είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και γι' αυτό στο τέλο τη ε, έκθεση μιλούμε για τη μελλοντική αλλαγή τη συνθήκη. και λέμε πώ θα πρέπει να γίνει αυτό. θα πρέπει να περιοριστούμε, να ασχοληθούμε μόνο σε ό,τι αφορά τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση ή να πούμε και σε άλλα ζητήματα μα απασχολούν. Αυτά είναι τα θέματα. Ε, αυτά αναφέρει και το γράφο και θέλουμε και τη δική σα άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τραρκόσκη, ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Το έγγραφο εργασίας για το οποίο ευχαριστώ τη γραμματεία της Επιτροπής μας η οποία το επεξεργάστηκε στην ουσία συγκεντρώνει και οργανώνει τα όσα έχουμε ετοιμάσεις αυτές τις εργασίες που ξεκινήσαμε πριν από κάποιους μήνες πλέον ε, για την πολυεπίπεδη εργασία. Ε, τα όσα κάναμε, η ακρόαση, ζητήσαμε και τη συνεισφορά από κάποιους συνταγματολόγους, ε, τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής μας στην έκθεση Tyson. Όλο αυτό το υλικό θεωρήσαμε ότι σιγά σιγά απέκτησε μια κάποια συνοχή και επομένως όλο αυτό που κάναμε εδώ, να οργανώσουμε όλο αυτό το υλικό, μας οδήγησε σε ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχει ένα ε, νήμα και επομένως μια βάση επί της οποίας θα ετοιμάσουμε ε, εμείς με τη σειρά μας ε, το σχέδιο έκθεσης. Βεβαίως ε, προκύπτουν ε, κάποιοι δεσμοί, κάποια ε, προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα τα λύσουμε και τι, πώς θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το οποίο κυριαρχεί, αν μου επιτρέπετε να συνοψίσω λίγο την κατάσταση, αφορά αυτή τη στιγμή θα έχουμε διευκρινίσει και καθορίσει το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία ανέκυψαν, παραδείγματο χάρη του πώς... Ε, Così, ε, la costruzione attuale θα ενσωματώσουμε το παρόν οικοδόμημα και θα του δώσουμε μια πιο συνεκτική εικόνα, διότι εμεί έχουμε κάποιε δομέ ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνηση που εντάσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο και κάποια εξωτερικά στοιχεία, κάποιου εξωτερικού οργανισμού και υπηρεσίε. και επομένω θα πρέπει να τα εντάξουμε όλα αυτά και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καθορίσουμε και να τροποποιήσουμε τι αρμοδιότητε αφενό και να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι διπλός λοιπόν ο στόχος ε, ένταξης και ανάπτυξης ε, που ε, από εκεί και πέρα άπτεται και μιας διπλής ανάγκης για συνεργασίας. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα, είναι οι, οι δύο διαφορετικές πτυχές του ίδιου νομίσματος και θα πρέπει να δούμε πώς το οικοδόμημα θα έχει ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα το έλλειμμα δημοκρατίας ε, ε, και το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας ε, πλήττει και την οικονομική διακυβέρνηση. Όλες αυτές λοιπόν οι απαιτήσει και όλοι αυτοί οι στόχοι μας οδηγούν σε κάποια διλήμματα, σε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι καταρχάς η ανάγκη να διατηρήσουμε αυτό το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να δημιουργήσουμε μια οικονομική και νομισματική ένωση ενισχυμένη στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, το οποίο αναπόφευκτα θα είναι πολύ ευρύτερο. Αυτή είναι η πρώτη ουσιαστική επιλογή που πρέπει να κάνουμε και αυτό θέλουμε να προτείνουμε και νομίζω ότι αυτή είναι και η βασική άγουσα ε, που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς αυτή την κατεύθυνση οδεύουν. Αυτό βέβαια είναι απλώς μια βάση. Στη συνέχεια το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα επιτύχουμε αυτό το διπλό στόχο της ένταξης και ανάπτυξης. Και εδώ θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό το μεταβατικό μοντέλο το οποίο σιγά σιγά έχουμε εκπονήσει. Δηλαδή να έχουμε μια διπλή τροχιά που θα είναι όμως δυναμική. Θα λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη αφενός και αφετέρου θα δούμε το θέμα της ε, μεταρρύθμισης των συνθήκων. Και εδώ φυσικά γίνεται και μια πολιτική εκτίμηση από πλευράς Κοινοβουλίου και από πλευράς της δικής μα της Επιτροπής σε σχέση με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία έχει πρόταση, πρόθεση να παρουσιάσει προτάσεις μεταρρύθμισης της συνθήκης πριν το τέλος της θητεία μα. Ε, βέβαια, εδώ η δική μα η έκθεση δεν είναι μια έκθεση η οποία μπορεί να προτείνει επισήμως μεταρρύθμιση των συνθήκων, αλλά ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να το συζητήσει η δική μας Επιτροπή ε, και να δούμε αν μπορούμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία μεταρρύθμισης των συνθήκων τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα μια επίσημη διαδικασία πρωτοβουλίας μεταρρύθμισης των συνθηκών από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα την ουσία των θεμάτων, Νομίζω ότι τα όσα έχουμε κάνει και τα οποία εν μέρη βασίζονται και στην έκθεση Tyson ε, εμβαθύνουν σε μεγάλο βαθμό ε, ως προς το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με βάση το παρόν νομικό πλαίσιο, που είναι πολλά αυτά που έχουμε να κάνουμε, το επαναλαμβάνω, αλλά φυσικά έχουμε αρκετή δουλειά ε, στην έκθεσή μας ε, στο μέτωπο αυτό, ιδίω όσον αφορά το θέμα της διαφοροποίησης των πόρων και όχι μόνο των κανόνων ε, στο παρονομικό πλαίσιο εδώ μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και νομίζω ότι αρχίζει να διαφαίνεται αυτό το οποίο είχαμε ως όρεμα ευθύ εξ αρχής, ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση στο παρονομικό πλαίσιο ε, μέσω των δύο διαφορετικών ε, δυνατοτήτων που έχουμε και στο fiscal capacity ε, προκύπτει κάτι το οποίο Ε, ουσιαστικά δέχεται την πρότασή μας στην έκθεση ε, Tyson να έχουμε αυτό το περιμερή προϋπολογισμό ε, στον προϋπολογισμό της Ένεσης και στο νομικό πλαίσιο. Μπορούμε βέβαια να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να περάσουμε σε πιο διεξοδική ανάλυση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε σήμερα, διότι πρέπει ε, να γίνει κατάλληλη συζήτηση γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να το θίξω, είναι η υποχρεώση του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόταση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ε, την οποία έχει εγκρίνει και η διάσκεψη των Προέδρων, υπάρχει και η συζήτηση εν εξελίξη για την ε, πιθανή σύσταση μιας υποεπιτροπής για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. θα πρέπει να είναι μια επιτροπή που θα είναι διαφορετική λόγω του αντικειμένου ή λόγω των μελών της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να ε, εκφράσει τις προτεραιότητές της και σίγουρα θα πρέπει να την απασχολήσει. Αναπόφευκτα λοιπόν το θέμα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στην έκθεσή μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της έκθεσης και πώς ε, συνδέεται αυτό στις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, πρέπει να πω ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αρκετά θετικά. Νομίζω ότι δέχτηκαν στο σημείο 14 των συμπερασμάτων τους ε, κάποιες ε, τροπολογίες ε, που είχαμε παρουσιάσει εμείς ως διαπραγματευτές εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Αυτή τις, αυτές τις έδρες της διακοινοβουλευτικής αντιπαρέθεσης θα έχουν δυνατότητες συζήτησης αλλά όχι ελέγχου. Και επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια το καθήκον να καθορίσουν πώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία, θα πρέπει και εμείς αναπόφευκτα να πούμε κάτι. Αν και νομίζω ότι θα σταθώ σε κάποιες αρχές και δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες για το σημείο αυτό. Ε, πέραν αυτού ε, υπάρχει, και το είπε και ο Ράφαλ, το πιο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τη φύση των πιθανών ε, ε, αλλαγών στη συνθήκη και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι πλέον προκύπτουν τρία μεγάλα μπλοκ στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Καταρχάς το θέμα των αρμοδιοτήτων, ιδίω ε, ως προς τον ορισμό, άρθρο 3.5 στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη φύση των αρμοδιοτήτων και το πώς κατανέμονται και από εκεί και πέρα ε, στα άρθρα για την, πολιτική, ε, για την οικονομική πολιτική πώς ε, ε, εντάσσονται αυτά. Υπάρχει και το θέμα της διαδικασίας και της ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πώς περνάμε λοιπόν στην πλήρη συναπόφαση και στη δυνατότητα για πλήρη συναπόφαση και υπάρχει και το τρίτο μπλοκ που είναι οι ε, χρηματοοικονομικές διατάξεις, ο προϋπολογισμός, οι διπόροι και σε αυτά τα τρία μπλοκ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ε, οδεύουν προς ποια κατεύθυνση και με αυτό ε, ολοκληρώνω. Όχι να κάνουμε το ομοσπονδιακό άλμα, αλλά προς μία μετάβαση ομοσπονδιακού τύπου, η οποία θα είναι σταδιακή και θα επιτρέπει μια δυνατότητα μιας πιο ήπιας ομοσπονδίας η οποία δεν θα θεωρείται ε, το τέλος, αλλά θα είναι το εφαλτήριο για μια συνέχεια την οποία θα καθορίσουν άλλοι και θα συνεισφέρουν και άλλοι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Κουαλτιέρη. Ο κύριος Ατερπέχη έχει το λόγο. Κυρία Γετρεπέχη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετική αυτή η έκθεση. Είναι μια διανοητική άσκηση, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου κάποια σημαντικά σημεία από πλευρά μου να σχολιάσω. Πάντοτε λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατή και ισχυρή όταν ε, κινείται ομαδικά, συνολικά. η εν τη ενός, αν θέλετε. Αυτό πραγματικά ε, ήταν η δύναμή μας τόσα χρόνια και αυτή τη γραμμή θα πρέπει να κρατήσουμε στο Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει ως σύνολο γιατί εκεί είναι και η πηγή της δύναμής μας. Πρέπει αυτό να το επισημάνουμε όσο γίνεται περισσότερο στον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας έχει αποδυναμωθεί η Επιτροπή και οι θέσεις της. Αν δούμε το παρελθόν, και τα συμπεράσματα συγκεκριμένα των τελευταίων δύο συνόδων κορυφής βλέπετε ότι ανατίθεται καθήκοντα στην Προεδρία του Συμβουλίου και στην Κομισιόν. Επ' αυτό πρέπει να τοποθετηθούμε και εμείς. Εμείς εμένουμε στη θέση του δικαίου πρωτοβουλία το έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θεωρούμε ότι είναι καλύτερη η διακυβερνητική προσέγγιση στα πράγματα. Έπειτα, η πιθανότητα Αλλαγή στο συνθήκων. Εγώ αυτό θα το συνέβαια με το άνοιγμα, με την ευελιξία. Οποιαδήποτε εξουσία να θέσουμε σε οποιαδήποτε επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτό δεν ε, χρειάζεται να αλλάξουν συνθήκε για να γίνει. Απαιτείται μάλλον πολιτική βούληση για να λαμβάνονται αποφάσει πιο ανοιχτά και να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν ε, τα τεκτενόμενα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρξε μία συζήτηση, συνεχή συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό όπως και για το ε, τις προσδομικές προοπτικές ε, της επόμενης περίοδου οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωβουλευτές, τα ΜΜΕ δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν ακριβώ τι συζητάτε στο Συμβούλιο, ούτε ποιε είναι οι προτάσεις οποιοδήποτε φορέα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε μια συζήτηση που γίνεται έτσι. Μπορούμε να δεχόμαστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τόσο κρίσιμα ζητήματα όπως είναι ο προπολογισμός στην επόμενη εφταετία χωρί χωρίς καμία διαφάνεια και πολλά άλλα ζητήματα που αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις ε, που ε, λαμβάνονται με πετροπολογία. μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν οι ψηφοφορίες γίνονται ανοιχτά και δημόσια, κανένα πρόβλημα. Αλλά η μυστική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και ιδίω η μυστικότητα ε, στη συζητήση για τον προπολογισμό είναι κάτι που δεν περιποιούν τιμή στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει το έγγραφό να επισημάνει το θέμα του ανοίγματο και της διαφάνειας. Κάτι άλλο που αφορά τη μέθοδο ψηφοφορίας εδώ στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές και την Ολομέλεια. Θυμηθείτε τη ψηφοφορία την περασμένη Πέμπτη. Πολλές φορές η ψηφοφορία είναι σαφής. 400 ψηφοί υπέρ, ε, και 200 κατά. Και βλέπουμε πολλέ φορέ ο πρόεδρο να λέει το αντίθετο. Πόσε φορέ ζητούμε έλεγχο ψηφοφορία. Λοιπόν, λάθη γίνονται. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά τα πράγματα θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα σήμερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε ε, το χέρι και ο πρόεδρος στο περίπου να κρίνει το αποτέλεσμα. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνεχώς και τα ε, λέμε και τα ξαναλέμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Μόνο αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να προβλέψουμε τα καθήκοντα και τον οποιοδήποτε. Και σε καμία περίπτωση ποτέ νωρίτερα. Πρέπει να υπάρχουν προποθέσει για την σωστή λειτουργία τη δημοκρατία.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 Το έγγραφο αυτό λέει πολύ συγκεκριμένα ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ε, αφορά μια μορφή διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ταχύτητες ε, ολοκλήρωσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι όλα τα κράτη έχουν την ομοθετική εξουσία, αλλά για κάποια θέματα, ιδίως για την Ευρωζώνη, ελάχιστα ε, μικρό, λιγότερα κράτη υπόκεινται στην ομοθεσία. Αυτοί λοιπόν που ε, δεν συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να έχουν και δικαίωμα να αποφασίσουν. Ο πρόεδρος ε, Σούλτς ε, στους Financial Times, νομίζω στις 7 Δεκεμβρίου, δεν είδα πουθενά άλλο αυτή την έκθεση, λέει ότι η, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να πάψει να είναι υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα, την Τραπεζική Ένωση και την Ευρωζώνη και αυτά θα πρέπει, συγγνώμη, η Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και αυτά θα πρέπει ε, να μεταφερθούν σε μια νέα επιτροπή που θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο. νομίζω ότι αναφέρθηκε ακροθυγός αυτό ο κύριος Γκουαλτιέρη, ελπίζω να κατάλαβα καλά. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτή είναι η προσωπική άποψη του κυρίου Σούλτ και μόνον ή αν αυτή η πρόταση έχει ευρύτερη ε, απήχηση. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές του Συμβουλίου και διαφορετικές εκδοχές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συνέχεια. Κάποιο να περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και κάποιο να περιλαμβάνει λιγότερα κράτη-μέλη. Η πρώτη μου αντίδραση στην πρόταση του κυρίου Σούλτς ήταν φυσικά ότι ενίσταμε στον αποκλεισμό των μελών της χώρας μου και ε, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι θα μπορούσε ίσως να είναι το πρώτο βήμα της αποκάλυψης του προγράμματος, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα προλιάνει το έδαφος για τη συζήτηση που πιστεύω ότι θα έρθει σίγουρα ε, την άνοιξη του 2015. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν την πολιτική συζήτηση για την ε, μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι επονίδιστο στο μεν, αλλά δυστυχώς, ε, συγγνώμη, ευτυχώς ε, παρέχει και τη δυνατότητα σε εμά να συμπληρώσουμε αυτό το κενό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται εδώ σε κρατέα θέση και μπορεί να καθοδηγήσει ε, το όλο θεματολόγιο της πολιτικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εξέπληξε το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο ζήτησε εμβάθυνση στη συζήτηση του θέματος στα κράτη-μέλη, αλλά δεν είπε τίποτα για το ρόλο των θεσμικών οργάνων στην όλη διαδικασία. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, σκοπεύει να δημοσιεύσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγή της συνθήκης την άνοιξη του 2014 που σημαίνει ότι θα είναι πολύ καθυστερημένες και δεν θα έχουν συνέπειες για την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δράσουμε γρήγορα προσεκτικά να επικεντρωθούμε στο θέμα της διακυβέρνησης πρωτίστως μιας ομοσπονδιακής οικονομικής διακυβέρνησης για τη Δημοσιονομική Ένωση και τι αυτό προϋποθέτει για τη δημοκρατία λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσε εξουσίες και δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Και να εξηγήσουμε και ποιο προφίλ αλλά και ποια μέσα θα πρέπει να έχει το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε την ε, Δημοσιονομική Ένωση καταλήλως. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο του έργου μας. Βεβαίως όλο αυτό θα επηρεάσει και όλα τα υπόλοιπα από την ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας μέχρι την ενία αγορά. Και θα πρέπει να περιλαμβάνει και απαραίτητος και το θέμα του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Πέραν της συμφωνίας η οποία επιτεύχθη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εικασίες για το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και η ίδια μια αναθεώρηση αρμοδιοτήτων, η οποία βαθμιδών θα ανακοινωθεί, θα υπάρξουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένη έρευνας, η οποία θα ολοκληρωθεί ε, στα τέλη του 2014. Ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Κάμερον, θα εκφωνήσει ένα λόγο τον Ιανουάριο, αυτό μας έχουν υποσχεθεί. Μας έχουν υποσχεθεί μία ε, μεγάλη ομιλία, η οποία θα διευκρινίσει τη στρατηγική και την τακτική του για το μέλλον των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να αντιληφθούν ότι οι σχέσεις της Βρετανίας αναδιαμορφώνονται ή ελοχεύει ο κίνδυνος να αναδιαμορφωθούν με διαφορετικούς όρους. Και φυσικά θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη ε, στην έκθεσή μας. Και τέλος, ε, μια τελευταία παρατήρηση, ε, μια τελευταία σκέψη για το Κοινοβούλιο. Βεβαίως και ρίζουν οι απόψεις στο Συμβούλιο και επαφίεται στο Συμβούλιο να αποφασίσει πώς θα διαμορφωθεί. Ε, αυτό είναι το όργανο το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Το Κοινοβούλιο όμως δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Και ο διαχωρισμός του Κοινοβουλίου σε επιτροπές οι οποίες θα αποκλείουν μέλη συγκεκριμένης εθνικότητας σίγουρα παραβιάζει τη συνθήκη και τον κανονισμό μας. Μπορεί λοιπόν κάλλιστα ο πρόεδρος Σούλτς και οποιοδήποτε άλλος ε, να εκφράζει τέτοιες ιδέες αλλά η Επιτροπή μας θα πρέπει να δώσει σαφή και ταχύτατη απάντηση ε, σε προτάσεις οι οποίες αν τεθούν σε εφαρμογή θα παραβιάζουν και τη συνθήκη και φυσικά θα μας εκθέσουν και θα μπορεί κάλλιστα κάποιο να τις αμφισβητήσει στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπροκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα Αυτά που είπε στο τέλος ο κύριος Σταφ για την νομική κατάσταση είναι σωστά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο βάσει της ε, ε, τωρινής συνθήκης μπορεί να πάρει γενική απόφαση. Δεν μπορεί να και δει δεν μπορεί να πάρθει απόφαση για το, προπολογισμό, για το προπολογισμό ή, αν δεν ε, ε, εμπλέκονται και τα 27 κράτη-μέλη. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο είναι όργανο της Ένωσης. Το είναι όμως και το Κοινοβούλιο του Ευρώ κατά συνέπεια. Είναι μια λογική συνέπεια η οποία είναι παιχνίδι λογικής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εξάγουμε τέτοιους συμπεράσματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή κάποια κράτη λένε ότι ε, κάποια κράτη-μέλη κάποια άλλα κράτη-μέλη ψηφίζουν και ψηφίζουν ε, μόνο και μόνο με τον τρόπο που ψηφίζουν, μόνο και μόνο επειδή δεν φύγονται αυτά τα ίδια. Δηλαδή τι κάνουμε, ότι ψηφίζουν κάποια κράτη-μέλη για να επιβληθούν σε άλλους πράγματα τα οποία δεν θα ήθελαν ποτέ να επιβληθούν στα ίδια αλλά επειδή δεν φύγονται τα ψηφίζουν. Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι γεγονός και είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Όταν συζητούμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, έρχεται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάνει μια ε, παρουσίαση ε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ο, ο πρόεδρος ας πούμε υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν εμφανίζονται εκεί μιλά, ε, γιατί λένε αυτό είναι θέμα της Ευρωζώνης δεν είναι θέμα δικό μας που είμαστε εκτός Ευρωζώνης Συγγνώμη ε, στο μέλλον θα έχουμε μια ευρωζώνη με όλο και περισσότερη Ευρώπη θα συζητιούνται τα πράγματα και θα αποφασίζονται και, από, δι' από ποιους από αυτούς που δεν θίγονται από τις αποφάσεις αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να προσέξει γιατί ε, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ποιοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις γιατί καταφέρουν θα καταλήξουμε σε παράλογα πράγματα Ευρωζώνη 17 μέλη θέλουμε ένα κοινοβούλιο 17 μελών όμως εγώ νομίζω ότι ο κύριος Βαν και ο πρόεδρος και ο κύριος Μπαρόζο και τα έγγραφά τους ε, ε, οδήγησαν τη συζήτηση σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλύτερη. Η ανησυχία είναι πως χωρίς να δημιουργήσουμε νομικό πρόβλημα θα δώσουμε το μήνυμα ότι βλέπουμε κάποια πράγματα ότι συνοδητοποιούμε ορισμένα πράγματα η συμπεριφορά του κοινοβουλίου η αυτορύθμιση αν θέλετε του κοινοβουλίου μπορεί να λειτουργήσει συμβολικά και να, να πούμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα κάποια πράγματα δεν γίναν σωστά αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πούμε ε, στους Βρετανούς φίλους μας να δώσουμε το μήνυμα ότι ναι μεν είπαμε ναι στην ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας και εγώ είμαι υπέρ αλλά εάν και εφόσον δεν θέλουν να έχουν παρτίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένα θέματα τουλάχιστον να μην ε, επηρεάζουν τις αποφάσεις και να μην ε, δημιουργούνται προβλήματα με τη συναπόφαση άμα κάτι δεν με ενδιαφέρει τον αφήνω στην ησυχία του το διπλανό μου δεν ξέρω είναι κάτι που κάνουν οι gentlemen νομίζω αυτό πρέπει να πούμε και από εκεί και πέρα μεταξύ μα αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Να αυτορυθμιζόμαστε εμεί, να αυτό περιοριζόμαστε και να συμπεριφερόμαστε ε, με τον σωστό τρόπο να πούμε ότι ορισμένα πράγματα ε, δεν έχουν σχέση με μένα είμαι gentleman ε, υπάρχει μεταξύ μας εδώ στο Κοινοβούλιο ένα gentleman's agreement να μην μένω στα χωράφια των αλωνών και να βάζω τρικλοποδιές για θέματα που τελικά δεν με αφορούν. Τι να σας πω τώρα. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να δημιουργούμε καινούρια κύματα, καινούρια τείχη στην Ευρώπη θα ήταν ντροπή νομίζω, θα ήταν κακό να α, κατακαιρματιστεί το κοινοβούλιο και τελικά να καταλήξουμε να λέμε ότι για ορισμένα θέματα ψηφίζει το κοινοβούλιο το 17, για άλλα θέματα ψηφίζει το κοινοβούλιο το 20, για άλλα το 27 κτλ. Κύριε Πρόγκ, ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα η παρεμβάση από δύο θέλουν να μας δώσουν κάποιο χρονοδιάγραμμα. Πότε θεωρείτε ότι θα είναι έτοιμο το σχέδιο γνωμοδότησης. Σήμερα ζητήσαμε ένα έγγραφο εργασία. Μόνο στα αγγλικά, ελπίζω σύντομα να έχουμε και μια μετάφραση στα ιταλικά και όχι μόνον. Για να μπορέσουμε να ξέσουμε καλύτερα τα κείμενα σα. Λοιπόν, τι προβλέπετε για το μέλλον, κύριε Γουαλτιέρη. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να πω και εγώ λίγα λόγια. Για τη συζήτηση που μόλις τώρα έγινε. Και για αυτή την πρόταση και υποποτρεπή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μπρόκ. Είμαστε ένα πολιτικό όργανο και θα πρέπει να φανούμε δυναμικοί και έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, όπου η σχολή σκέψης εκείνη που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δομικά δεν μπορεί να αποτελέσει, να επιτελέσει μάλλον τον ρόλο ενός πραγματικού Ευρωκοινοβουλίου της Ευρωζώνης, τότε η μόνη λύση είναι η διακυβερνητική λύση. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τις συνθήκες. Οι συνθήκες είναι η βάση μας. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί στη στάση μας. Πιστεύω ότι έχουμε και επιτυχίες. Και θέλω να πω ότι στο επίπεδο της ε, δημοκρατικής νομοποίησης, το συμπεράσμα του Συμβουλίου λέει κάτι πολύ ε, θετικό για μας δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα και να υπάρξει αυτή η δήλωση και πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή του ίδιου του Προέδρου, μια πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ καλά ετέθη ως πρωτοβουλία Για να έχει λοιπόν αυτή η πρόταση για να δείξει τη σημασία του ζητήματος και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ιδίως σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Και για να μπω στην ουσία του θέματος, εγώ δεν θεωρώ και θα ήμουν κατά, αν θέλετε, σε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν πιστεύω λοιπόν θα υπάρξει μια λύση τέτοια που η... επισημοποιεί, αν θέλετε, τη διακριτική μεταχείριση κάποιων συναδέλφων μέσω μιας υποεπιτροπής. Αντίθετα, θεωρούμε ότι όπως υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας που είναι διαφορετική από την ε, ευρωπαϊκή πολιτική, ε, εξωτερική πολιτική ε, και υπάρχουν λοιπόν και διαφορετικά όργανα που ασχολούνται με αυτές τις δύο πολιτικές θα μπορούσαμε να έχουμε μια υποεπιτροπή που να εμβαθύνει σε θέματα ευρωζώνης πάντα μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Και όπως εχει οπτάει ότι η Δανία για την ε, πολιτική άμυνας και ασφάλεια. πώς αυτό μεταφράζεται, ότι δεν υπάρχουν μέλη, τακτικά μέλη στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Μόνο ένα αναπληρωματικό μέλος. Όχι ότι απαγορεύεται να είναι οι άνθρωποι μέλη, αλλά είναι κοινή λογική. Η λογική που ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Μπροκ. Αυτό θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε, μια λύση, μια επιθυμητή λύση, ώστε να διασφαλίσουμε την ισότητα όλων των συναδέλφων, όλων των μελών, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και ένα σαφές και ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή και είναι ικανό να αντιμετωπίσει ε, ενστάσεις και ερωτηματικά σχετικά με την ομιμότητα που το καλύπτει αν ε, ασχοληθεί περαιτέρω με θέματα ευρωζώνης. στο μέλλον θα υπάρξει περαιτέρω διαφοροποίηση που να βασίζεται και, στους πόρους και όχι μόνο στους κανόνες, μπορεί να υπάρξει. Άρα πράγματι αυτό ενισχύει και τη θέση ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσαρμοστεί. Τώρα καταλήξουμε να έχουμε συνεδριάσεις ε, αν θέλετε, για θέματα ευρωπαϊκού υπολογισμού που να συμμετέχουν μέλη μόνο από κάποια μέλη, δεν είναι επιθυμητό. Θα πρέπει όμως το Κοινοβούλιο ως νομοθέτης να διασφαλίσει τα προνόμια που έχει. Αυτό που απλά θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα και να προετοιμαστούμε για τη μελλοντική αυτή συζήτηση όπως θα δημορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Τώρα πιο συγκεκριμένα για το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι καλά κάναμε και περιμέναμε. Τώρα έχουν τεθεί στο τραπέζι για κάποιες προτάσεις και συμφωνώ με τον κύριο Νταφ. Η καταληκτική ημερομηνία που εδόθη για την Επιτροπή είναι πολύ μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν χρονικό ορίζοντα που να μας επιτρέπει να κλείσουμε αυτή την έκθεση έγκαιρα, ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσει μια δική του πρόταση πριν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το όριο για μένα. Μέσα σε αυτό το όριο και επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέβαλε έως τον Ιούνιο την υποβολή αυτού του δικού χάρτη για τον οικονομικό και δημοσιονομικό πυλώνα, ε, ας επωφεληθούμε κι εμείς για να έχουμε τον επαρκή και κατάλληλο χρόνο, ώστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη συζήτηση και με την κατάλληλη δυναμική. Τι εννοώ, δεν χρειάζεται να βιαστούμε περιβολικά όσο το Γενάρη να έχουμε ήδη ένα σχέδιο ε, έκθεσης και να κλείσουμε γρήγορα αυτή την άσκηση. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ως χρονικό ορίζοντα το επόμενο εξάμεινο. <coughs> Οπότε ίσως το Φλεβάρι, εντάξει, να το συζητήσουμε. Κάπου το Φλεβάρι να υπάρξει ένα σχέδιο λοιπόν κειμένου, ώστε ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Ιούνι να μπορεί να το συζητήσει το Κοινοβούλιο, να τοποθετηθεί ε, γενικός προσανατολισμός είναι αυτός που λέω. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό πιο συγκεκριμένο το επόμενο διάστημα. Ε, Κύριε Ταρκόφσκι, θέλετε να προσθέσετε κάτι κι εσείς. Ε, όχι, σας καλύπτει ο συνάδελφος. Καλώς. Κλείνει το μικρόφωνο του Προέδρου. Πρέπει να ορίσουμε ημερομηνία εκ νέου για την συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. 18 Φεβρουαρίου λοιπόν είναι η επόμενη ημερομηνία συζήτησης. Αυτή είναι η απόφασή μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο που πάλι αφορά τους δύο συζητητές, τους κυρίους Ρακόφσκι και Βαλτιέρη. Η έκθεση αυτή αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των εκλογών του 2014. Η διάσκεψη των Προέδρων επιβεβαίωσε τη δυνατότητα να έχουμε και πάλι δύο εισηγητές. Προχωρούμε λοιπόν γιατί το άρθρο 14 παράγραφος 2 της συνθήκης μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ας ακούσουμε τις απόψεις των δύο συνεισυχητών. Κύριε Γουαλτιέρ. Uh, Ευχαριστώ. As you know, in... Όπως γνωρίζετε, το 2014 το επόμενο κοινοβούλιο έχει ένα καθεστώς εξαίρεσης ε, το οποίο ισχύει τώρα για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, το οποίο λύγει για την επόμενη θητεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διπλή εξαίρεση, διπλή παρέκκληση στην ε, ε, διάταξη της συνθήκης για την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια παρέκκληση που μας επιτρέπει, επιτρέπει να διατηρήσουμε 99 έδρες αντί των 96 ως μέγιστο ανώτατο όριο. Επομένως έχουμε Συγγνώμη, η γερμανική καμπίνα λέει ότι έχετε δύο μικρόφωνα ανοιχτά και παρενοχλείτε ε, το μικρόφωνο του ομιλητή. Και υπάρχει και μια δεύτερη παρέκκληση για την Κροατία που θα επιτρέπει να γίνουν οι 12 Κροάτες παρατηρητές ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλέον των 754 μελών που έχουμε αυτή τη στιγμή Επομένως, το Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της αιτίας του, όταν θα ολοκληρωθεί το θέμα της προσχώρησης της Κροατίας, θα έχει 766 έδρες. Επομένως, πρέπει για την επόμενη θητεία από τους 766 να περάσουμε στους 751, διότι θα λήξει το καθεστώς παρέκκλησης, εκτός ε, και αν γίνει αλλαγή της συνθήκης, κάτι το οποίο είναι απίθανο. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τη σύνθεση του Κοινοβουλίου στις διατάξεις της συνθήκης βάσει μιας διαδικασίας που είναι η διαδικασία του άρθρου 14.2 της συνθήκης το οποίο προβλέπει ότι μέσω πρότασης του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου, με τη συνένεση και πάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω, είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση. για μια σύνθεση η οποία θα σέβεται τον αριθμό των 7, 750 ε, βουλευτών συν τον πρόεδρο ε, και έτσι να έχουμε τα δύο ελάχιστα και μέγιστα ανώτατα όρια, 6 και 96 βουλευτές. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης ε, ε, πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να μπορέσει και να μεταφραστεί το κείμενο και νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τρεις αρχές τις οποίες θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Η πρώτη είναι το θέμα της ε, ε, βαθμιδών μειούμενης αναλογικότητας, η οποία είναι μια πολύ σημαντική ε, αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, διότι είμαστε μια ένωση πολιτών και κρατών μελών και θα πρέπει να εξισορροπούμε και την εκπροσώπηση των πολιτών βάσει της αρχής ένας άνθρωπος μία ψήφος και Μία αρχή που διέπει όλα τα ομοσπονδιακά κράτη για την εκπροσώπηση των κρατών μελών. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας όπως ορίστηκε στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης Λαμασούρ Σεβερίν λέει ότι όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός ε, τόσο μεγαλύτερο το δικαίωμα να αυξηθεί ο αριθμός των εδρών και επίσης δεύτερον όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός τόσο περισσότεροι πολίτες θα εκπροσωπούνται από το κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, η οποία είναι μια αρχή. Δεν μπορούμε να την ε, ε, ε, ξεχνούμε, διότι τεχνικώς είναι αδύνατο να τηρήσουμε αυτό το 100%. Το να γίνει πλήρως σεβαστό to have the same number ε, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να έχει τον ίδιο αριθμό εδρών. Είναι λοιπόν μια τεχνική διάταξη, ε, από αυτή την άποψη δεν είναι πολιτική, αλλά είναι μια αρχή την οποία πρέπει να σεβαστούμε, πρέπει να διασφαλίσουμε την αναλογικότητα, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε και αυτή τη φθήνουσα διαδικασία. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι κάτι το οποίο αναφέρεται επίση στην έκθεση Σεβερίν Λαμασούρ, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρω ε, τα ελάχιστα και μέγιστα όρια, διότι δεν είναι υποχρέωση. Ε, το 96 είναι το μέγιστο όριο, δεν είναι όμω υποχρέωση. Και από πολιτική όμως σκοπιά και για θεσμικούς λόγους θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο αναλογικότητας. Και αυτό έχει ως σαφή συνέπεια ότι αν θέλουμε να σεβαστούμε το μέγιστο όριο και να ακολουθήσουμε και την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, θεωρητικά θα πρέπει, για παράδειγμα, να αυξήσουμε τις έδρες της Γαλλίας, διότι αλλιώς θα πρέπει να μειώσουμε τις έδρες της Γερμανίας ή να μην σεβαστούμε την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας αλλά όπως σας είπα, εδώ αναφερόμαστε σε μία αρχή που διέπει τις αποφάσεις μας, αλλά όχι μία πλήρη υποχρέωση. Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη καταρχάς την ευθύνουσα ε, διαδικασία και κατά δεύτερον την αναλογικότητα. Και για να χρησιμοποιήσουμε τα μέγιστα όρια που διαθέτουμε και επίσης διότι γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση της Λισαβόνας στο Γερμανικό Σταγματικό Δικαστήριο αναφέρθηκε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετή αναλογικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήττει την ομιμάτωτά του. Εγώ είμαι κατάφορα αντίθετο σε αυτό το επιχείρημα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει συγκεκριμένη ένσταση και δεν μπορούμε και πάλι ε, να... Ε, ε, περάσουμε πέραν το ορίου από όσο γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι Εάν δούμε τις ιστορικές αλλαγές των θέσεων από το 1979 των εδρών ε, μέχρι σήμερα, είναι σαφές ότι έχουμε ε, πειράξει λίγο τη φθήνουσα αναλογικότητα σε σχέση με το πώ είναι η κατάσταση και οι μεγάλε χώρε έχουν χάσει πολύ περισσότερε ε, έδρε από τι μεσαίου μεγέθου και τι μικρότερε. και επομένω αυτό το μέγιστο όριο είναι το μέγιστο. Δεν μπορούμε να πάμε πέραν από αυτόν διότι δάλο ε, το όλο θέμα τη ε, νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ε, αμφισβητηθεί ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο λοιπόν εδώ, το οποίο θα πρέπει να μεταφραστεί σε κάποιο μαθηματικό τύπο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια μεγάλη ανακατανομή. Αν ε, δούμε για παράδειγμα τα δύο βασικά μοντέλα, το μοντέλο του Cambridge και το παραβολικό μοντέλο, στο μοντέλο του Cambridge υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανακατανομή η οποία δεν νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη. Και αν λάβουμε υπόψη και το φθήνοντα ρόλο του μαθηματικού τύπου χρησιμοποιώντας το παραβολικό μοντέλο, εκεί θα δούμε ότι δεν αρκεί μόνο να μειώσουμε τις έδρες για να βρούμε αρκετές έδρες για την Κροατία, αλλά θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ανακατανομή για να γίνουν σεβαστές οι δύο πρώτες αρχές. Και εδώ φτάνουμε στο τρίτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, που είναι η κοινή λογική. Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για να ε, σεβαστούμε τη φθήνουσα αναλογικότητα και το ανώτερο όριο θα πρέπει να γίνει μια τόσο μεγάλη ανακατανομή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και μια τρίτη αρχή που είναι ο ρεαλισμός, η κοινή λογική και το γεγονός ότι αυτή η διάταξη και αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα. Επομένως, θεωρώ, και αυτό είναι και το καταληκτικό μου επιχείρημα, ότι θα πρέπει να προτείνουμε μία ρεαλιστική λύση, όπως την αποκαλώ. Η ρεαλιστική λύση θα λάβει υπόψη την ανάγκη της φθήνουσας αναλογικότητας και την ανάγκη να υπάρχει αρκετή αναλογικότητα προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το μέγιστο όριο και να μην ε, ε, μας παρουσιάσει και πάλι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας ε, θέματα που αμφισβήτησης της νομιμοποίησής μας και να χρησιμοποιήσουμε μια ρεαλιστική λύση η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρότασή μας θα πρέπει να είναι μια πρόταση που θα είναι ένα πάρε δώσε. Δεν κερδίζει κανεί έδρες, αλλά και κανείς δεν θα πρέπει να χάσει πάνω από μία. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός μας προσανατολισμός. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τα δύο πρώτα στοιχεία στον απαραίτητο ρεαλισμό για να υπάρχει ευρύτερη συνένεση στο Κοινοβούλιο και επίσης για να είναι πιο πιθανή η ομόφωνη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να παρουσιάσουμε συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά να ξέρετε ότι και αυτό το επεξεργαζόμαστε. Αλλά αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να παρουσιάσουμε εδώ στην Επιτροπή μας την αρχή που θα διέπει την πρότασή μας, που είναι η αρχή μιας λύσης που θα λάβει υπόψη και την ανάγκη της φθήνουσας αναλογικότητας, αλλά και την ανάγκη για ρεαλισμό. I think that I can stop here. Θα σταματήσω εδώ. Ωραία λοιπόν. Έχω πολλούς ε, εγγεγραμμένους ομιλητές. Καταρχάς όμως ο κύριος Σταρκόφσκι. Well, I, I just to say... Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ε, κάποια γενικά σχόλια και να απευθύνω και κάποιες γενικές ευχαριστίες. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και είναι δύσκολο πραγματικά να μιλούμε για θέμα τέτοιων εδρών του Κοινοβουλίου. Είχαμε κάποιε άτυπε επαφέ για αυτό το ζήτημα και ακόμα και μία έδρα να χαθεί για οποιοδήποτε κράτο μέλο είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί οποιοδήποτε ε, και το γνωρίζουμε. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που βάλουμε στο τραπέζι την πιο πρακτική και ρεαλιστική λύση που μπορεί κανείς να φανταστεί μακάρι να φτάσουμε στην κατάσταση εκείνη όπου κανένα κράτο μέλο να μην χάσει παραπάνω από μία έδρα. Αλλά να είμαι ειλικρινή, αυτό δεν είναι δίκαιο και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Αν καταλήξουμε σε μια τέτοια ρεαλιστική λύση, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πραγματικά εναλλακτική. Η μόνη άλλη εναλλακτική θα ήταν να ζητήσουμε αύξηση των εδρών του Κοινοβουλίου συνολικά. Δηλαδή, η μόνη άλλη εναλλακτική είναι να πούμε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και η μόνη πρότασή μας είναι να ζητήσουμε επιπρόσθετες 12 έδρες. Και δεν θέλω καν να πάω σε αυτή τη λύση, γιατί φανταστείτε τι εικόνα θα δώσει το Κοινοβούλιο σε μια εποχή κρίσης. το μόνο που κάνει το Κοινοβούλιο είναι να αυξάνει τις έδρες του. Γνωρίζω βεβαίως απόλυτα ότι είναι αδύνατο να κάνουμε μια επαναστατική ελεγγύη στο Κοινοβούλιο χωρίς ταυτόχρονα να συντηθούν και άλλα ε, θεσμικά ζητήματα όπως είναι η ψήφη στο Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εξίσου ρεαλιστές. Ιδανική λύση δεν υπάρχει και στο μέλλον θα συζητούμε τη μελλοντική συνθήκη, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα και να βρούμε μια πιο ριζοσπαστική λύση. Πάντως, το πλέον σημαντικό είναι και πολύ ορθά το είπε ο Ρομπέρτο, που μίλησε για το περιεχόμενο διαφόρων προτάσεων που ακούστηκαν. Γιατί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο γίνονται οι προτάσεις. Για μας το πιο σημαντικό θέμα είναι ε, ο ορισμός Λαμασούρ για την ε, αναλογικότητα ε, με φθήνουσα τάση. Στην τελευταία θητεία αυτό ψήφισε και ε, το Κοινοβούλιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε την αναλογία ανάμεσα στον πληθυσμό και τις έντρες. Και θα πρέπει λοιπόν εφόσον ακολουθούμε μια φθήνουσα πορεία από Γερμανία έως την Μάλτα και το Λουξεμβούργο να λαμβάνουμε υπόψη ε, τον πληθυσμό. Ας αφήσουμε οποιοδήποτε μαθηματικό, μαθηματικό τύπο στην άκρη. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να λάβουμε υπόψη μόνο τις ιστορικές εξελίξεις ε, και την ε, κυρίαρχη αρχή του ε, Λαμασού, τότε θα πρέπει κάποια κρατημέλη να αυξήσουν κατά δύο-τρεις έδρες την, τις έδρες και αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη τις δημοκρατικές τάσεις, κάποιοι θα πρέπει να χάσουν τρεις έδρες και παραπάνω. Πάντως όλοι τουλάχιστον μία έδρα. Αν λοιπόν θέλουμε να πάμε παραπέρα και να αποδεχτούμε αυτό τον κανόνα, το κανόνα δεν είναι εύκολο, κάποια κράτη-μέλη να κερδίσουν κάποιε έδρε και να ξέρουν ότι στο μέλλον μπορεί με την εκβάθρον αλλαγή τη συνθήκη αυτό να αλλάξει, τότε θα πρέπει α, να γίνει αυτό. Ιδάλω θα πρέπει να μειώσουμε τι έδρε τη Κροατία. Αλλιώ θα εφαρμόσουμε αυστηρά την αρχή Λαμασόρ σχετικά με την απόλυτη αναλογία, αυστηρή αναλογία ανάμεσα στον πληθυσμό και τις έδρες. Δεν το κάνουμε με αυτό. Γιατί πολιτικά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποδεχτούν τα κράτη-μέλη που θίγονται. Γιατί κάποιοι λένε α, χάνουμε μία-δύο έδρες α, χωρίς να γίνεται συνολικά μια διαπραγμάτευση για όλους. προτείνουμε κάποιοι προτείνουμε κάποιοι να χάσουν μία έδρα. Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες αποκλήσεις ε, στη λύση προτείνουμε. Γιατί είπα και πριν, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, κάποιοι πρέπει να χάσουν δύο έδρες. βάζουμε αυτή την στο τραπέζι χωρίς να θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν και τίποτα μη ρελιστικό. Το αντίθετο. Απλά θέλω να σας πω ότι πολύ απλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Η εναλλακτική θα ήταν να ζητήσει το κοινοβούλιο σε μια τόσο δύσκολη χρονική στιγμή επιπρόσθετε έδρες. Θεωρώ ότι αυτό είναι διανόητο. Αδιανόητο και για μας, ε, στην Επιτροπή μας, αλλά γενικότερα για το Κοινοβούλιο. Αν πραγματικά μας νοιάζει η εικόνα του Κοινοβουλίου και αν θέλουμε να κοιτάμε και στο μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις στο μέλλον και θέλουμε εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να διαπραγματευτούμε πιο ουσιαστικές αλλαγές, θα πρέπει να κρατήσουμε μια πιο ψυχρεμη στάση. Ο κύριος Νταφ. Uh, we begin... Ξαναρχίζει το ίδιο βιολί Πάντως εγώ θα ήθελα να τονίσω το κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος αυτού. Η ένταξη της Κροατίας έχει οριστεί για τον Ιούλιο. Οι Κροάτες θα έχουν ένα κάποιο αριθμό ευρωβουλευτών, 11 συγκεκριμένα, αν σας ενδιαφέρει βέβαια. Και είχαμε συμφωνήσει ότι καλύτερο θα ήταν να έχει πάρθει η τελική απόφαση μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Αυτό ήταν ο στόχος μας για να συμφωνήσουμε για τις έδρες στο επόμενο κοινοβουλίο, στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί το δικαίωμα του να πάρει πρωτοβουλία για ένα θέμα σαν και αυτό λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας που μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε, ας το κάνουμε σωστά. Ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η όλη διαδικασία θα πάει καλύτερα από το παζάρι και το αλυσβερίσι ανατολικού τύπου που κάναμε στο παρελθόν. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πακέτο αν θέλετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο αλυσβερίσι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια γραμμή του προπολογισμού για να μετριάσουμε τον πόνο εκείνης της χώρας που χάνει μια έδρα. Άρα τα πράγματα θα είναι ο δύσκολα για να καταλήξουμε. Στο κοινοβούλιο αυτό θα Έχουμε δυσκολίες λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες. Βεβαίως προς το παρόν ε, δρούμε κατά παράβαση της συνθήκης. Η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας δεν τηρείται με την ε, σύνθεση αυτή τη στιγμή του Κοινοβουλίου. Ο Ρομπέρτο βέβαια αυτή τη ρήτρα την ονόμασε προσανατολισμό γενικό αλλά εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και νομικό κριτήριο και από ό,τι γνωρίζω το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρεί την αρχή της ευθύνουσας αναλογικότητας και την τήρησή της ως νομικό κριτήριο και όχι απλά γραμμή προσανατολιστική. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να παραλύσουμε από την γραμμή Λαμασούρ Σεβερίν πέρασε από το κοινοβούλιο το θέμα αυτό αλλά δεν μπήκε σε κανένα νομικό κείμενο αυτό γι' αυτό ξανά προτείνω όπως έχω πει και στο παρελθόν τροποποίησε αυτής της φόρμουλας Λαμασούρα Σεβερίν. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα λογικό και διαφανές συμπέρασμα. Γιατί ό,τι απόφαση πάρουμε θα πρέπει να την εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας. Να τους εξηγήσουμε γιατί γίνεται κατανομή των εδρών έτσι όπως γίνεται. Μέχρι τώρα δεν τα είχαμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό ποτέ. Ας το κάνουμε τώρα. Βεβαίως η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, θα πρέπει να, να συμφωνηθεί και η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ε, νομική φόρμουλα αν θέλετε σε ένα νομικό κειμενάκι που θα πρέπει να προστεθεί σε οποιαδήποτε συνθήκη μας διέπει. Φαντάζομαι ότι τον, την άνοιξη θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση η οποία να ανατρέψει αν θέλετε αυτά που ισχύουν τώρα. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειές μας και Ε, θα, αν θέλουμε να πούμε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα χάσει πάνω από μια έδρα τότε αναζητούμε 11 κράτη-μέλη ως εθελοντές που είναι πρόθυμα να χάσουν μια έδρα, έναν ευρωβουλευτή. Τώρα κάποια κράτη-μέλη θεωρούν τους ευρωβουλευτές πιο σημαντικούς από ό,τι τους θεωρούν άλλα. Με μεγάλη περιέργεια περιμένω να δω ποιοι θα είναι οι εθελοντές οι οποίοι θα αναλάβουν να χάσουν μια έδρα ο καθένας. Σοβαρό όντως αυτό το θέμα. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Ρομπέρτο και τον Ραφαέλ για την παρουσίασή τους. Χαίρομαι που κανείς τους δεν θέλει να μεγαλώσει τον αριθμό των βουλευτών του Κοινοβουλίου. 754 είναι κάμποση. Ε, και εγώ θα έλεγα κιόλα στόχος μας είναι το 751. Τώρα βέβαια στο Συμβούλιο η πρόταση φαίνεται να ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα λοιπόν αν προτείνουμε εμείς μια αρχική πρόταση κάτω από 751 μπορεί να μην ξεπεράσουμε πολύ το, ε, το νούμερο που θα θέλαμε. Τώρα μία έδρα να χάσει ο γιατί όχι δύο αν, επειδή πρόκειται και για διαπραγματεύσεις, αν ξεκινήσουμε με 750, 751 έδρες, με 11 ε, ε, maximum απώλειες αυτό δεν είναι ουσιαστικά διαπραγμάτευση είναι αυτή η τελική μας θέση αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο λοιπόν εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε μείον τις τρεις γερμανικές θέσεις ε, και μία από κάθε κράτος μέλος άρα μείον 30 7.36 λοιπόν αρχίζουμε με την πρόταση για μια μικρότερη λοιπόν ε, μικρότερη σύνθεση του κοινοβουλίου εξοικονομούμε ε, και λεφτά του φορολογουμένου αλλά αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία χάνει τρεις έδρες και μετά ε, θέλουμε και μια χώρα να χάσει ο καθένας ε, από τους υπόλοιπους όπως είπε και ο Νταφ ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι εθελοντές ένα λεπτό πρόεδρε ένα λεπτό πρόεδρε μια τεχνική διευκρίνηση θέλω να κάνω γιατί έχω την εντύπωση ότι παίρνει μια τροπή η συζήτηση που είναι λανθασμένη από νομική διευκρίνηση πρώτον τι λέει η συνθήκη. Η συνθήκη λέει δεν θα παζαρέψουμε το μέγεθος του κοινοβουλίου. 751 έδρας. 751 έδρας. Αυτό είναι. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Άρα δεν υπάρχει. Ε, δεν υπάρχουν αλλαγές. Τέλειωσε. Δεν αρχίζουμε λοιπόν διαπραγματεύσεις για το μέγεθος του Κοινοβουλίου. Ούτε να τα αυξήσουμε τις έδρες μπορούμε, ούτε να τις μειώσουμε. Οπότε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε πρόταση με 751 έδρες. Εκεί τελειώνει. Το Συμβούλιο ψηφίζει με ομοφωνία. Το Κοινοβούλιο συνενεί. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο δεν κάνει διαπραγματεύσεις. Εμείς θα πούμε ειδού η πρότασή μας θα συνενέσουμε άμα σεβαστείτε την πρότασή μας. Διαπραγματεύσεις δεν κάνουμε και ιδιαίτερα, αυτή είναι η νομική κατάσταση. Ιδιαίτερα για το μέγεθος του Κοινοβουλίου. Άγνιο. Εγώ προέρχομαι από την ανατολική περιφέρεια του Ηνωμένου Βασιλείου 5,5 εκατομμύρια πολίτες 7 ευρωβουλευτές έχουμε στην Κύπρο ο πληθυσμός είναι 1 εκατομμύριο και έχουν 6 ευρωβουλευτές είναι τεράστια η στρέβλωση εδώ Επιπλέον υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Τα 5,5 εκατομμύρια του Ηνωμένου Βασιλείου της περιοχής μου ε, είναι καθαρή συνεισφορίες ενώ στην Κύπρο απλώς παίρνουν hear what he said, sorry. Σχόλιο εκτός μικροφώνου Right, apparently the objection to increasing the size of the house Φαίνεται ότι η αντίρρηση για την να μεγαλώσουμε το μέγεθος του κοινοβουλίου είναι οικονομική. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι άμα θέλετε υπερ αντιπροσώπευση τότε πληρώστε. Άμα οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν, να βάλουν, να μετρήσουμε ας πούμε πόσο κοστίζει ο ευρωβουλευτής και να πούμε ότι δίκαιο είναι άμα θέλετε παραπάνω ευρωβουλευτές να ψηφί, πληρώσουν οι πολίτες. Ήδη από την αρχή της συζήτησης ε, είχα εκπλαγεί. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω πώς ο συνάδελφος Φόξ να θεωρεί ότι 751 έδρες είναι υπερβολικά τόσες πολλές για 450 εκατομμύρια πολίτες. Σκεφτείτε πόσε έδρε έχετε στη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων. Ε, πρώτα απ' όλα πάτε και τακτοποιήστε τα του οίκου σα και μετά λέτε και να τα, μας τα ξαναπείτε αυτά. Εκτός μικροφώνου κάποια σχόλια. Δεν μιλάω σε εσά, μιλώ ε, στην άδεια καρέκλα του κυρίου Φόξ. Έτσι δεν είναι. Απλά είσαστε δίπλα. Τι να κάνουμε. είναι το μόνο που μπορώ να είπω. Δεν απευθύνθηκα όμω σε γιατί δεν πήρατε εσεί το λόγο. Επίτα, ο συνάδελφος ο κύριος Νταφ ε, εντυπωσιάζει με τα επιχειρήματά του. Καταφέρνει πραγματικά να μιλάει για το ζήτημα χωρίς να αναφέρεται στο Συμβούλιο. Πώς προτείνει κανείς δηλαδή να αλλάξει η ισορροπία στο Κοινοβούλιο χωρίς ούτε μία κουβέντα να κάνει για το Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία εδώ στο Κοινοβούλιο, χωρίς να αλλάξει η ισορροπία στο Συμβούλιο. Πραγματικά κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική στο Συμβούλιο. Το Σύνταγμα της Γερμανίας προβλέπεται 49 και από την άλλη Βλέπουμε πώς γίνεται κατανομή ανάμεσα στα διάφορα κρατήδια. Έξι ψήφοι, για παράδειγμα, στη Βεσφαλία. Αν δώσουμε τρεις ψήφους στην Κύπρο και τρεις στο, στη Γερμανία, σκεφτείτε την πολύ αυστηρή αναλογία που θα υπάρξει. Αλλά δεν είναι κανείς που το δεχτεί. Όχι, διαφωνών. Και δεν καταλήγουν σε κανέναν κανόνα στο Συμβούλιο, αλλά θέλουν να επιβάλλουν κανόνα στο Κοινοβούλιο. θέλουν να έχουν μια διπλή εκπροσώπηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και λένε από τη μία δημογραφικά κριτήρια και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αδύνατο όμως αυτό. Τη μέρα που θα δεχτείτε να αντιμετωπίσετε ισότιμα τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, τουλάχιστον με έναν λογικό τρόπο, αν όχι ισότιμο, ε, τότε, τότε, να μιλήσετε και για αναλογικότητα στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό. Διότι θέλετε ισότητα των πληθυσμών, αλλά όχι ισότητα των κρατών. Δείτε τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, στην Ελβετία, την Βραζιλία, το Μεξικό, την Ινδία. Δηλαδή θέλετε κράτη πρώτης ταχύτητας και κράτη δεύτερης ταχύτητας και και ομοσπονδία στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό. Ποιοι είναι λοιπόν οι φεντρελιστές τελικά αυτοί που κάνουν διαφοροποιήσεις ε, στο ανώτερο σώμα ή αυτοί που θέλουν να κρατήσουν διαφορές και στο ανώτερο και στην άνω και στην κάτω βουλή. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Εμείς μπορούμε να σεβαστούμε απόλυτα την αρχή της ευθύνους αναλογικότητας και να δεχτούμε την πρότασή σας για την Κροατία. Όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στα μεγάλα κράτη, θα πρέπει να κάνουν μια διευθέτηση ανάμεσα Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Να κάνουν μια διευθέτηση μεταξύ τους και να κάνετε κάποιες αλλαγές. Και θα καταλήξετε στην φθηνούς αναλογικότητα. Για τους πολύ καλά μας έχει αποδείξει ο Λαμάσορ, αν χάσει κάποιε έτερες η Γερμανία τότε και η Γαλλία δεν θέλει διαθέσει από σήμερα. Θα πρέπει να θυσιαστούν τελικά οι μεσαίες χώρες για να εφαρμόσουμε απόλυτα την ιδέα της φθήνωσης αναλογικότητας. Αυτό που λέω είναι ότι η πρόταση που ακούσαμε από τους δύο συγγητές είναι επικοδομητική πρόταση. Ρεαλιστική και επικοδομητική. Διαφωνώ όμως με τη βάση του επιχειρήματος. Αν θέλετε μια ομοσπονδία, πάντοτε θα πρέπει να έχουν, αν θέλετε, ε, αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και πώς λειτουργούμε με την άνω Βουλή. και αν δέχεστε ω κριτήριο το δημογραφικό στοιχείο στο κοινοβούλιο δεν μπορείτε να το αποκλείετε α, στο ε, κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση των μέσων, μεσαίων και μικρών κρατών. Αυτό είναι ατύπημα που πρέπει να το πληρώσουμε όλοι. Αν δεν υπάρχει συμμεταχείριση, επαναλαμβάνω, στο Συμβούλιο. Δεν είναι αντιδημοκρατικό λοιπόν αυτό. Ούτε καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα περί μη δημοκρατικού χαρακτήρα. Ενώ κάποιοι να, να κρίνεται ένα μάλλον αποτέλεσμα στι εκλογέ με 3-5%. Αυτό είναι δημοκρατικό. Και αυτό που λέμε τώρα εδώ είναι αντιδημοκρατικό. Κοιτάξτε, αυτό που σημαίνει δηλαδή στη Βρετανία είναι πολύ διαφορετικό. Οι περιφέρειε εκλογέ στη Βρετανία είναι πολύ διαφορετικέ. Σε κάποιε περιφέρειε εκλέγεται μόνο έναν βουλευτή με πολύ μικρό εκλογικό σώμα, ενώ σε άλλε περιφέρειε είναι πολύ μεγάλο το εκλογικό σώμα. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει στην Ευρώπη συμβαίνει και στην ε, Βρετανία. Δεν είναι τόσο διαφορετικό το πράγμα. Και μάλιστα σε περιπτώσει στη χώρα σα είχε κάτι χειρότερο. Λοιπόν, δημοκρατία είναι το κράτο δικαίου. Και είναι και ένα πάζλ. Είναι ένα μεικτό σύνταγμα, όπως μας δίδαξε ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αν δεν θέλετε μια ισορροπημένη λύση, ε, τότε θα πρέπει οι μεσαίες χώρες θα είναι κατά αυτές τις λύσεις και δεν πρόκειται να περάσει από το Συμβούλιο αυτή η πρόταση. Και λέω, δεν είπα ότι διαφωνώ με την πρόταση και, τη λογική των ε, δύο συγκητών, γιατί είναι πολύ ρευστική λύση. Αυτό που δεν μπορώ όμω να δεχτώ σε καμία περίπτωση και που πολλέ χώρε που είναι ακριβώ αυτή τη μεσαία κατηγορία δεν πρόκειται να δεχτούν, είναι αυτό το επιχείρημα που απευθύνεται. Γιατί είναι πραγματικά υποκριτικό επιχείρημα. Όμω, Μάλλον φεντεραλιστές να είμαστε, μεν, αλλά κάποια κράτη-μέλη είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους, αν θέλετε. Σε ένα φεντεραλιστικό οικοδόμημα δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια επιχειρήματα. Χρειαζόμαστε λύσεις που να βασίζονται σε κάποιες γενικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιαδενμάκη. Σας ευχαριστώ. Οι πολίτες φαντάζονται ότι η κατανομή εδώ καθορίζεται με μαθηματικό τύπο. Φαντάζομαι όμως ότι θα πρέπει να ε, ακούσουν τη συζήτησή μας εδώ για να καταλάβουν ότι είναι πολύ περισσότερο από έναν απλό μαθηματικό τύπο και μάλιστα το ζήτημα είναι ιδιαίτερα καυτό. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, αυτή η φθήνουσα αναλογικότητα, η οποία μέχρι τούδε γίνεται σεβαστή. Έχουμε την έκθεση Λαμασούρ Σεβερίν, η οποία δικαίως ε, χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αρχή. Επίσης αναφερθήκαμε στη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται στη συνθήκη και ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω όμως ότι ε, κανονικά θα έπρεπε με να αυξήσουμε την ε, ε, σύνθεση του Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ποσά. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε την αρχή της φθήνης ως αναλογικότητας. Σας ευχαριστούμε γιατί ήσασταν και σύντομοι και σαφείς. Ο κύριος Χέφνερ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές πως σε αυτήν την ε, συζήτηση μπαίνουν ουσιαστικά θέματα πολύ βασικά της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κτλ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σωστά για να φτάσουμε σε σαφή αποτελέσματα. Εγώ αυτή την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας δεν ότι θεωρώ ε, απαραίτητη δεν είναι επαρκής κατά την απόψή μου μπήκε στις συνθήκες βέβαια αλλά είναι ο λίγον τι ευσεβής πόθος η αρχή αυτή από την οποία συνεχώς αποκλίνουμε εγώ νομίζω ότι η αρχή αυτή είναι μπορεί να είναι από νομική άποψη αρχή αλλά θα πρέπει να τηρείται 100% τότε γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε κάποιους κανόνες Κάποιους κανόνες μπορούν να εφαρμαστούν 100%. Η δικαιοσύνη, η θέμης στην αρχαία Ελλάδα έχει κλειστά τα μάτια. Λοιπόν και εμείς θα πρέπει να βρούμε κανόνες εδώ που με κλειστά τα μάτια να μπορούμε να τους εφαρμόζουμε. Να θα πρέπει να ξεφύγουμε από διαδικασίες που λέει υποτίθεται ότι αναφέρονται σε μια κάποια αρχή αλλά ουσιαστικά η μόνη αρχή που τις διέπει είναι η αυθαιρεσία όποιος θέλει ακολουθεί την αρχή όποιος θέλει δεν την ακολουθεί λοιπόν αυτό δυστυχώς είναι έτσι γι' αυτό εγώ λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε τι φιλοδοξία να καταλήξουμε εδώ σε μια φόρμουλα, σε κάποιους κανόνες που να, μπορεί, να μπορούν να εφαρμοστούν ούτω ώστε να μην αρχίσουμε, αρχίζουμε με κάθε καινούργια προσχώρηση στο μέλλον να α, κουβεντιάζουμε επί μήνες πώς, ποιος είναι ο αριθμός των νέων βουλευτών κτλ. Να πω ότι Τώρα κύριε Άγνιου αυτό που είπατε με τρόμαξε. Ήτανε πλακά. Αστείο ήτανε ή ήταν πραγματική πρόταση. Για να είμαι ειλικρινής, το να αγοράζει ο πολίτης έδρες στο κοινοβούλιο είναι, τι να σας πω, σηκώνεται η τρίχα. Ε, έχουμε ακούσει πολλά πράγματα βέβαια από εσά. Έχουμε και διαφορετική άποψη για το ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο πολίτης, ποια είναι η δημοκρατία. Αλλά τόσο εξωφρενικό πράγμα δεν είχα ξανακούσει από εσά. Τώρα, για τον Ραφαέλ, τον Αντζέλ. Συγγνώμη, αναφερθήκατε στο γερμανικό σύνταγμα αναφερθήκατε σε αυτό και είπατε ότι στην, στο Bundesrat είναι διαφορετική σύνθεση από ότι είναι στο Bundestag. Τα μεγέθη που είναι κάπως διαφορετικά. Ωραία. Να σας πω όμως ότι εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ ποτέ να πάρτε σαν μοντέλο το γερμανικό σύνταγμα και στο Bundesrat το συνταγματικό δικαστήριο στην Καλσρούι αναφέρθηκε στο Bundesrat και είπε one man one vote τώρα αν θέλετε εσείς one member state one vote άλλος ο λογαριασμός ε, έτσι ε, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια κάποια ισορροπία ε, δεν ε, είναι τα πράγματα τόσο τρομερά όσο υπονοήσατε σε αυτά που είπατε ε, ότι επελέγει δηλαδή στο Συμβούλιο κάτι το οποίο βρωμάει λίγο, δεν, είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν θέλετε να φανταστείτε βέβαια ο, ένα σύστημα με δύο βουλές, τότε μπορούσατε να πάρετε ε, το σύνταγμα με σαν μοντέλο αν και πάλι δεν θα ήταν σωστό όπως είπε και ο συνάδελφος υπάρχουν ορισμένα πράγματα από τα οποία, τα οποία είναι δεδομένα. 751 είναι το νούμερο και η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας είναι και αυτή δεδομένη. Συζητήσαμε ήδη δυο μοντέλα εδώ στην Επιτροπή όταν κουβεντιάζαμε την αλλαγή του εκλογικού συστήματος και την έννοια της εκλογικής περιφέρειας για τις ευρωπαϊκές εκλογές και λέω ότι η αρχή αυτή αν θέλουμε μάλλον να, εφαρμόσουμε αυτή την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας χωρίς τεράστιες ανατροπές στο νούμερο των εδρών Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να γίνει από όσο το δυνατόν περισσότερους αποδεκτό αυτό το μοντέλο που θα φτιάξουμε και για μένα η φόρμουλα είναι παραβολική. Παραβολική, δηλαδή βαθμιαία με την αύξηση του πληθυσμού αυξάνεται και ο αριθμός των δωρών αλλά η έδρα αναλογεί σε περισσότερα άτομα. Επουδενή λόγο θεωρώ ότι μπορούμε να δεχθούμε γραμμική αύξηση, παραβολική πρέπει να είναι όπως σας είπα, ε, διότι με τη γραμμική αύξηση θα είχαμε τεράστια προβλήματα, ούτε ο συμβιβασμό του Κέμπριτζ δεν μπορώ να δεχθώ αλλά όλα αυτά τα άλλα μοντέλα είναι όλα αυθαίρετα. Δεν και δεν θα περνούσαν σε κανένα συνταγματικό δικαστήριο τελικά μεταξύ μας. Γι' αυτό λέω ας βρούμε μια λύση η οποία και από τον κόσμο να μπορεί να γίνει αποδεκτή αλλά και από το Συμβούλιο και από από τα δικαστήρια λοιπά Τώρα, όσον αφορά τα, τη φόρμουλα την παραβολική, εγώ έκανα διάφορους υπολογισμούς. Έτσι γιατί από μαθηματική άποψη δεν υπάρχει μία φόρμουλα μόνο παραβολική, υπάρχουν πολλές. Λοιπόν, Προσπάθησα να δω τι γίνεται και με μεγάλη χαρά θα κουβέντιαζα όλους αυτούς τους πιθανούς υπολογισμούς. Κάντε τους κι εσείς γιατί πρέπει να φτάσουμε νομίζω σε μία λύση η οποία μπορεί να είναι ρεαλιστική αλλά να είναι και λιγάκι διαχρονική να, να, ζήσει για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι αυτές που είχαμε βρει μέχρι τώρα. Παρόλα. Ωραία, ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω είναι πάντα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μεταρρυθμίσει στον φορέα στον οποίο ανήκει. Ζητούμε μεταρρυθμίσει από όλα τα άλλα όργανα, αλλά το δικό μας το όργανο να το μεταρρυθμίσουμε μας πέφτει δύσκολο. Είναι γεγονός αυτό. Όμως χρειάζεται μεταρρύθμιση στο δικό μας το όργανο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα είμαστε κλωτσοσκούφοι των κυβερνήσεων και για τις έδρες και για το, τον αριθμό των εδρών και ε, για την κατανομή των εδρών. Αυτό δεν τα, αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. Δεν τα αποφασίζει δυστυχώς μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχά... Ε, έκτοτε βέβαια, τώρα όμω πρόσφατα μάλλον, υπάρχει η Λισαβόνα και το, η δοκιμή της Λισαβόνας δεν θα πρέπει να, την, να αποτύχουμε σε αυτήν. Αν δούμε ιστορικά τι έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο αριθμό των Ευρωβουλευτών, θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα πρώτα ότι ξεκίνησε ως συμβουλευτικό όργανο το κοινοβούλιο έκτοτε γίναμε νομοθετικό όργανο και εξελισσόμαστε σε, και ένα όργανο με, νομοθετική και δημοσ, με νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες ωστόσο η αντιπροσωπευτικότητα πρέπει να ε, διατηρηθεί και τώρα φτάνει η Κροατία και εδώ πρέπει να πάρουμε απόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η φθήνους αναλογικότητα περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι βασική νομική αρχή και θα ξέρω αν θυμάστε στη συνέλευση προσπαθούσαμε να κάνουμε, να βρούμε μια αντίστοιχη ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου δεν έπεσε από τον ουρανό ε, έγιναν τεράστιες συζητήσεις και βρέθηκε και μια συμβιβαστική λύση η οποία είναι ο λίγο της για την Ευρωπαϊκή Ένωση διπλή πλειοψηφία για το Συμβούλιο και α, φθήνους αναλογικότητα για το Κοινοβούλιο. Ε, κύριε συνάδελφοι υπάρχουν πολλά συστήματα με δύο βουλές τι να σας πω διαφορετικά όμως λειτουργούν οι δύο ε, οι δύο βουλές ε, στις χώρες που τις έχουν. Στη Γερμανία έχουμε από Σάρλαντ, έχουμε μοναχά ε, τρεις ψήφους του Nordline Westfalen έχει έξι. Ωραία, αυτή, αυτή ήταν μια συνένεση που βρέθηκε μετά τον πόλεμο, έτσι. Το, στη Γερμανία του 48 ε, ε γίνανε κάποιες ε, παραχωρήσεις έτσι ε, τέλος πάντων είναι σου η λύση στη Γερμανία ενώ υπάρχουν άλλες χώρες ε, όπου ε, δουλεύουν διαφορετικά υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα και εν πάση περιπτώσει εδώ να συνειδητοποιήσουμε και όλα ότι δεν μιλάμε για συνθήκη μιλάμε για πρωτόκολλο που θέλουμε να αλλάξουμε τώρα έτσι Λοιπόν, είναι δεδομένο μας λέει και είναι αλήθεια αυτό η φθήνουσα αναλογικότητα. Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε ένα μαθηματικό τύπο, μια φόρμουλα που να ε, μας βολεύει όχι μόνο για την ένταξη της Κροατίας αλλά και για τις επόμενες προχωρήσεις, ξε, προσχωρήσεις, ξέρω εγώ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο δεν είμαι μάγος, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά στην συνέλευση είχαμε πει ότι υπάρχει ένα ελάχιστο νούμερο 4. Το Λουξεμβούργο είχε 6 έδρες και ο Ζαν Κλοντ γιουμκερ ήταν πολύ σημαντικός εκείνη την εποχή, ε. λάβετε το υπόψη σας. Τώρα πια το Λουξεμβούργο δεν είναι και τόσο σημαντικό. Έχουμε, τη, ε, έχουμε και τη Μάλτα που είναι πιο μικρή από το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία είναι πιο μικρή. Έχουμε 5-6 Λουξεμβούργα δηλαδή όσον αφορά το μέγεθος. Ε, και τελικά μία έδρα αντιπροσωπεύει 60.000 άτομα από τη Μάλτα αλλά 800.000 από ένα μεγάλο κράτος μέλος εντάξει δεν πειράζει δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ ε, Τέλος πάντων, μακάρι να βρούμε μια λύση με μεγάλη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Διότι άμα έχουμε πολύ μικρή πλειοψηφία εδώ, δεν θα επιβιώσει η πρότασή μας στο Συμβούλιο. Ε. Θέλουμε μεγάλη πλειοψηφία. Αυτά είχα να πω. Ωραία, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Πολύ σοβαρή. Ο κύριος Λεγκρίπ. Η, η κυρία Λεγκρίπ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν λεχθεί πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Απλά να τονίσω αυτά που είπαν οι δύο συνεισηγητές. Ήταν σωστά, ρεαλιστικά. Περμένω βέβαια και τις επόμενες συζητήσεις μετά από τη σημερινή πολύ βασική συζήτηση που αναφέρθηκε σε βασικές δημοκρατικές αρχές, ισορροπίες κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο, μιας και έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, Κάπου τα περιθώρια μας είναι περιορισμένα. Ε, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Είναι η Κροατία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να έρθουν σε μας οι Κροατοί ευρωβουλευτές. Να βρούμε έναν τρόπο να τους υποδεχθούμε, να δείξουμε μια κάποια φαντασία, μια κάποια δημιουργικότητα, ωστόσο να κάνουμε κάτι που να μπορεί τελικά να θεωρηθεί να είναι δηλαδή, στο να, κάνουμε, να βρούμε μια λύση που να είναι α, πραγματικά στο επίπεδο του κοινοβουλίου που θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω. Ας α, ε, παραμείνουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο που έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ας α, ε, δούμε και την αρχή τώρα η φόρμουλα Λαμασούρ Σεβερίν δεν εφαρμόζεται όπως μας είπαν ακούστηκε η μάξιμο απώλεια μιας έδρας ε, που πρέπει να γίνει σεβαστή. Ας σεβαστούμε λοιπόν τις συνθήκες. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Και ας μην μπούμε στον πειρασμό να προτείνουμε πράγματα όπως τους κάνει αύξηση του αριθμού του μεγέθους του κοινοβουλίου. Του χρόνου έχουμε εκλογέ. Μα ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν η λύση που θα βρούμε να είναι ε, άξια του κοινοβουλίου μα απέναντι στην κοινή. Ευχαριστώ κυρία Γεννάκου. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα δεν είναι απλώς τεχνικό, είναι βαθιά πολιτικό θέμα όπως γνωρίζουμε η κατανομή των εδρών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και οι αποφάσεις στο κορεπέρ έχουν μια ιδιαιτερότητα που θέλει τις μικρές και τις μεγάλες χώρες να έχουν μια ισορροπία μεταξύ τους ώστε να μην απειλείται το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένος πολιτικός λόγος. Άρα ούτε η πλήρης αναλογική, ούτε οι μαθηματικές φόρμουλες, ούτε αυτά μπορούν να θεραπεύσουν μια τέτοια κατάσταση και οι συνεχείς αλλαγές βέβαια στην ε, ε, σύνθεση του Κοινοβουλίου ε, μπορούν να επιφέρουν και απαιτήσει των κρατών μερών για αλλαγές στο επίπεδο του Κορεπέρ. Διότι δεν είναι δυνατόν να ανατρέπεται μόνο το Κοινοβούλιο. Ε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που υπάρχει να αλλάξει ο αριθμός του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να αφαιρεθούν έδρες. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε τι έγινε στην τελευταία διεύρυνση. Αφαιρέθηκαν έδρες από ορισμένε χώρες. Ας πούμε από τη χώρα μου αφαιρέθηκαν τρεις έδρες. Επομένω υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή αν αφαιρέθει μια έδρα. Διότι συμπαθής είναι η προσέγγιση όσων δεν τους αγγίζει το θέμα γιατί σε τελευταία ανάλυση κάποιος θα πρέπει να απαντήσει στο εσωτερικό της χώρας γιατί αφαιρέθηκαν οι έδρες από αυτές τις χώρες και όχι από άλλες. Επομένως το θέμα, όπως είπε και ο κύριος Ζανζέλ, δεν είναι τόσο απλό. Βεβαίως θα αποφασιστεί στο Συμβούλιο, αλλά η γνώμη του Κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία. Και νομίζω ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να μεταβάλλεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ούτε πρέπει, μπορεί να έρχονται συνεχώς νέες απαιτήσει για το πώς θα είναι η σύνθεση του Κοινοβουλίου. Διότι τότε αλλάζει ο ρόλος του και εφόσον αλλάζει ο ρόλος του αλλάζει και η πολιτική ουσία για την οποία έγινε Δημοκρατικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννάκου. Ο κύριος Βίλαντ. Ähm, Ευχαριστώ. Μετά θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Χέφνερ. Κύριε Ραντζέλ, όλα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, που είπατε, είναι από εθνικής απόψεως σωστά. Αλλά από ευρωπαϊκή σκοπιά δεν είναι σωστά. Λέτε, αν είχαμε δύο βουλές σαν ε, όπως έχει η Γερμανία θα έπρεπε να κάνω αυτό ναι αλλά πάρτε τότε και το πρώτο και το, την πρώτη βουλή έχουμε πλήρη αναλογικότητα στην άλλη βουλή έτσι δεν ισχύουν αυτά που ισχύουν στο Bundesrat λοιπόν και σας, σας λέω οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό φαντάζομαι ούτε από εσά, έτσι λοιπόν τέλος πάντων κυρίες και κύριοι πριν από την μεγάλη ένταξη των 10 και νέων χωρών μελών το 2004 είχαμε πει ότι θέλουμε 700 βουλευτές και εγώ θεωρώ ότι 700 είναι καλοί. Κάποιος είπε ότι είναι ένας, μια προσανατολιστική καθοδή ε, καθοδηγητική γραμμή ε, το 751 ε, η οποία εφαρμόζεται ως προσανατολισμός όχι τυφλά κυρία Γιαννάκου α, ως προσανατολισμός από εκεί και πέρα το σημαντικό σημείο είναι ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο κανόνα. Μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει αν αύριο το κάποιο κράτος μέλος στην απογραφή που θα κάνει έχει 20% παραπάνω μεγαλύτερο πληθυσμό ή κάποιο άλλο κράτος μέλος έχει 30% χαμηλότερο πληθυσμό Μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει λοιπόν αν, αν τα πράγματα αλλάξουν σε επόμενες εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Και κυρία Λεγκρίπ, ακριβώς το πλεονέκτημα του να αποφασίσουμε ήδη από τώρα για μια διαχρονική φόρμουλα είναι ακριβώς για να αποφύγουμε να έχουμε τέτοιου είδους εκνευριστικές συζητήσεις στο παραπέντε μέσα σε ένα κλίμα πανικού, πανικού στην επόμενη προσχώρηση. Δεν γιατί σας λέω ότι αν δεν πάρουμε τη σωστή απόφαση τώρα θα ξαναλέμε τα ίδια πράγματα στο μέλλον. Ας βρούμε ένα κανόνα, όπως είπε και ο συνάδελφος Λάνεν, που να μπορεί να εφαρμοστεί διαχρονικά και ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το κανόνα αυτό σωστά, σωστά. Ε, κοιτάξτε, τώρα βέβαια μπορείτε να... Ε, ε, το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτά που θα αποφασίζουμε τώρα θα πρέπει να μπορούν να ε, εφαρμοστούν στο μέλλον. Βέβαια σε 15 χρόνια δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ίδια ακρίβεια και ούτε κανείς θα σας πυροβολήσει επειδή βάλατε την υπογραφή σας σε αυτό εδώ. Τι να σας πω. Ε, τώρα από εκεί και πέρα αν εφαρμόζονται, αν εφαρμόζονται ε, οι κανόνες που αποφασίζουμε ε, σωστά ε, δεν είμαστε παιδάκια του σχολείου νομίζω ότι βλέπουμε όλοι τι θα έπρεπε να γίνεται και δεν γίνεται και θα μπορούσαμε να πούμε να χάσουν δύο έδρες από κάθε χώρα αλλά αν κάποια χώρα έχει κάτω από το 10% του συλλογικού ευρωπαϊκού πληθυσμού να μην μπορεί να χάσει δύο έδρες, να χάσει μοναχά μία ακόμη και αν υπολογίζει θα έπρεπε να χάσει παραπάνω ε, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν, κάνουμε τους υπολογισμού μας μέχρι το 29, διότι μετά το 2029 ο Δής γνωρίζει αν θα υπάρχει ο κόσμος. Ε. Ευχαριστώ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ε, και έχουμε ακόμα μια παρέμβαση. Έχει ζητήσει το λόγο να απαντήσει και ο κύριος Ρανζίλ. Πρώτα η κυρία Τάιλ και μετά ο κύριος Ρανζέλ, αλλά πρακτικά πολύ συνεπτική. Ευχαριστώ συμφωνούμε νομίζω τουλάχιστον ότι το μάξιμο μόριο είναι 751 και εγώ ασχολήθηκα με τους μαθηματικούς τύπους και είδα ότι πολλές από αυτές τις μαθηματικές φόρμουλες καθοδηγούνται ουσιαστικά από εθνικά συμφέροντα οπότε σε τελευταία ανάλυση μπορούμε ε, μπορούμε να αποκλείσουμε τις ε, άλλες φόρμουλες να παραμείνουμε στην παραβολική η οποία όμως και αυτή μπορεί να αλλάξει από 750 έως 759 θα ε, ο Γερμανός πολίτης όμως επειδή είναι το σύνταγμά μας αυτό που είναι δεν μπορεί να δεχθεί θεωρεί ότι είναι αδικό αυτό που λέμε ότι ε, ότι δεν υπάρχει στη Γερμανία one man one vote σε όλα τα επίπεδα. Ε, ξέρω ότι πάρθηκαν α, αποφάσεις την περασμένη φορά ας πούμε ήταν ε, έγινε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 ε, υπάρξει συζητήσεις και αποφάσεις οι οποίες τελικά θα οδηγούσαν αν θέλετε σε ε, ε μείωση του αριθμού των φιλελευθέρων ε, έχουμε έξι ε, ευρωβουλευτές εμείς ε, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε μείωση του αριθμού. Εγώ είμαι η πρώτη φιλελεύθερη ευρωβουλευτή από το Βερολίνο και προσωπώ 5,5 εκατομμύρια. Τώρα ο Βρετανός συνάδελφος δεν είναι εδώ για να ε, τα ακούσει αυτά που λέω. Έχετε την εντύπωση ότι είμαι πολύ, το, είμαι επιπλέον, ε, θα μπορούσα να φύγω να μην υπάρχω εδώ. Και έκανα και μια άλλη δουλειά πέρα από τον υπολογισμό το, με τους μαθηματικούς τύπους ε, είδα ότι 14 ευρωβουλευτές δεν έρχονται καν. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Wenn alle wirklich mitarbeiten würden, ja, also so da wären, wie sie eigentlich dazu verpflichtet sind. Λοιπόν, λέω ότι αν όλοι εδώ στο αυτό το κοινοβούλιο δούλευαν όπως έπρεπε να δουλέψουν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Τη Μαρίν Λεπέν δεν την είδα εδώ. Αν δουλεύαμε όμως όλοι καλά δεν χρειαζόμαστε ούτε 751. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο πρόεδρος ζητά λίγη υπομονή ε, επιπλέον ε, στους διερμηνείς για να μιλήσουν οι κύριοι Ρανζέλ και ο κύριος Γουαλτιέρη, αλλά πραγματικά συνοπτικά. Πολύ σύντομα, τεχνικά διαδικαστικό προς τον κύριο Βίλαντ, διότι είπε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά αναλογικά το εκλογικό σύστημα της Γερμανίας και αυτό δεν ισχύει, διότι με το, με μεικτό εκλογικό σύστημα μπορούμε να εκλέξουμε ανθρώπους που δεν θα έλαμβαναν έδρα αν είχαμε μόνο τον κανόνα της αναλογικότητας και στην γερμανική κυβέρνηση δίνεται μία λύση, προστίθενται κάποια μέλη για να ε, αναπληρώσουν ε, το ονομαστικά αναλογικό σύστημα. Δεν είναι μόνο αυστηρά αναλογικό. Συζήτηση εκτός μικροφώνου με τον κύριο Βίλαντ. Δεν είναι πραγματικό αναλογικό, επιμένει ο κύριος Ράνχελ. Έχετε ένα μαθηματικό τύπο, αλλά δεν είναι αναλογικός. Δεν είναι, επιμένει ο κύριος Ράγχελ. Σας το ε, διαβεβαιώ και μπορώ και να σας το αποδείξω. Η βασική αρχή είναι η αναλογικότητα, απαντά ο κύριος Βίλαντ, και μόνο όταν έχουμε ερετά μέλη. Μπορεί να συμβεί όμως να υπάρχει κάποιος ε, ο οποίος ε, λείπει. Ο πρόεδρος, σας παρακαλώ μην διακόπτετε το ένα στον άλλον. Μια δεύτερη παρατήρηση, ο κύριος Ράγχελ, διότι έχω δει πολλούς που κατάλαβαν τι ε, εννοεί ο κύριος Γκουαλτιέρη, θα σας το πει και ο ίδιος, με τη βασική αρχή. Η αρχή είναι ένα νομικό κριτήριο. Είναι ένα κριτήριο το οποίο απορρέει από τον νόμο, αλλά δεν είναι κανόνας, δεν είναι ακριβής κανόνας. Και εσείς που είστε Γερμανοί και έχετε σπουδάσει δίκαιο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η γερμανική θεωρία ε, της ε, νομοθεσίας έχει τις δύο αυτές βασικές αρχές, τις αρχές και τους νόμους και τους κανόνες. Και τι λέει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ότι δίνουμε μια πολιτική κατεύθυνση, δεν είναι πολιτική κατεύθυνση με την έννοια της ε, αγγλικής, του αγγλοσαξονικού δικαίου, αλλά είναι μια αρχή ε, βάσει της οποίας δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό είναι σαφές. Σας προτείνω να διαβάσετε το μέτρο τελειέρα Πρόεδρος, ωραία. Πριν δώσω το λόγο στους κύριου Σταρκόφσκι και Γκουαλτιέρη, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει από τους δύο, ο κύριος Σταρκόφσκι φαντάζομαι εκ μέρους του κυρίου Γκουαλτιέρη επίσης, επειδή αρχίζουν και φεύγουν και οι συνάδελφοι, να σας πω λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα συζητηθεί το θέμα αυτό, λογικά στις 21 Ιανουαρίου, θα υπάρχει, ελπίζω, ένα σχέδιο έξιδεθεσης, αυτό καθ' αυτό. Ο κύριος Σταρκόφσκι, για να ολοκληρώσουμε. Ήθελα απλώ να πω ότι ή θα πρέπει να γίνει ένα καδικαμαικό σεμινάριο ή κάποια μέλη θα πρέπει να φύγουν για καφέ και να καθυστερήσει αυτός ο καφές ιδιαίτερα να διαρκέσει πολύ. Δεν μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας όλες, είναι δύσκολες ερωτήσεις. Αν ε, θέλουμε να ανατρέψουμε τελείως το σύστημα το οποίο θέλουμε να επιλέξουμε θα πρέπει να γίνει εν μέσω σύμβασης και από εκεί και πέρα θα ληφθούν απόψη, υπόψη όλες οι θέσεις των ε, κρατών μελών και των ε, ευρωβουλευτών. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό το ζέσταμα που κάναμε εδώ. Πρέπει να σκεφτούμε μια ρεαλιστική λύση και του χρόνου να σκεφτούμε κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να προτείνουμε ε, στο Συμβούλιο χωρίς να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Ε, σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Πρέπει να αποχωρήσω δυστυχώς. Ο Πρόεδρος. Κύριε Γκουαλτιέρη, ολοκληρώστε εσείς. Θα παρουσιάσουμε την έκθεση τρία πράγματα να πω διευκρινιστικά. Πρώτον, οι ισορροπίες στην αντιπροσώπευση στα θεσμικά όργανα είναι ιστορικής φύσεως που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ο καθένας έχει την ιστορία του και δεν μπορούμε από εκεί και πέρα να έχουμε μία ε, προσέγγιση μιμητική. Σε κάθε χώρα υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που αποτελούν τμήμα ε, μιας ζωντανής διαμόρφωσης. Και συμφωνώ με τον κύριο Ράγκελ ότι υπάρχει και η φθήνουσα αναλογικότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε. Τελεία και πέβλα. Είναι μια αρχή όπως σας είπα διότι δεν μπορεί από τεχνική σκοπιάς διότι έχουμε δύο αρχές. Κάθε κράτος για να έχει περισσότερες έδρες, εάν το σεβαστούμε αυτό, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο χώρες με τον ίδιο αριθμό εδρών. Ήδη αυτό από μόνο του λοιπόν αποδεικνύει ότι μιλάμε για μια αρχή και όχι για ένα κανόνα, όπως έλεγε δικαίως ο κύριος ε, Ράγκε. Είναι όμως μια αρχή η οποία ισχύει και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την τηρήσουμε. Δεύτερον, είναι σαφές ότι δεν έχουμε ένα Αμυγό αναλογικό σύστημα στο Συμβούλιο και δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να γίνει γερουσία. Στο Συμβούλιο υπάρχει το θέμα της ομοφωνίας, υπάρχει και η ρήτρα ε, για την ε, ε, στενή προσέγγιση με, το, με τον πληθυσμό, είναι φθήνουσα διαδικασία. Δεν πρέπει να έχουμε αμυγό αναλογικό σύστημα, είναι κάτι το οποίο είναι αναλογικό μεν, αλλά με κάποιες αποχρώσεις. Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι μπορούμε να κάνουμε καταμερισμούς, αναδιακλαδώσεις και οι μεγάλοι να τα βρούνε μεταξύ τους. Διότι ακριβώς λόγω της έκθεσης Λαμασούρ Σεβερίν αυτό θα μείωνε τους βουλευτές της Γερμανίας και ο Λαμασούρ λέει σαφώς ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ψαλίδα πλήρως. Επομένως δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ε, την υπόθεση να μειώσουμε τη Γερμανία κάτω από τους 96 διότι ήδη ε, είναι αρκετά λίγοι οι βουλευτές της και αναπόφευκτα θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη λύση που θα πρέπει να έχει ή ένα προσανατολισμό και εδώ συμφωνώ με το Βίλαντ ή μια κατεύθυνση και εγώ συμφωνώ με το παραβολικό μοντέλο αλλά δεν μπορεί εδώ τώρα να ε, αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον παραβολικό τύπο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές και να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο ε, όπου δεν αυξάνονται οι έδρες, δεν μειώνονται σε κανέναν οι έδρες περισσότερο από μία και χρησιμοποιούμε να, εξακολουθούμε να τηρούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε κανόνα 100% για τους λόγους που σας εξήγησα. Ευχαριστώ, ε, ωραία σας ευχαριστώ όλους για μια θερμή και διεξοδική συζήτηση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς ο Πρόεδρος. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτέ, καλά Χριστούγεννα και να σκεφτείτε ακόμα περισσότερο τα θέματα αυτά. Ευχές σε όλους.